Καλησπέρα σε όλους σας. Uh, Είναι η πρώτη επίσημη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού στην οποία προεδρεύω και πολύ περήφανος είμαι που βρίσκομαι εδώ. Και τα επόμενα, το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια και μήνες ελπίζω να έχουμε γόνιμη συνεργασία με καλές αποφάσεις. will that. Έτσι, ώστε όλοι να καταλάβουν ότι είμαστε εδώ και δουλεύουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ημερήσια διάταξη. Σας ενημερώνω ότι τα σημεία 9 και 17 έχουν αλλάξει μεταξύ τους. Φυσικά αυτό δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία των θεμάτων, όπως καταλαβαίνετε. Και στη συνέχεια θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Ελπίζω να συμφωνείτε με αυτή τη μικρή αλλαγή στη μερίσια διάταξη. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι το ε, τελευταίος διάλογος τριμερής για το προσχέδιο προϋπολογισμών 2020 θα λάβει χώρα στο Συμβούλιο αύριο στις 23 Ιουλίου. Αυτή ήταν η τελευταία ανακοίνωση και φτάσαμε ήδη στο σημείο 3. Εάν προχωρήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα αυτή την ταχύτητα θα τα ξεπετάξουμε όλα, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα γίνει. Το 3. Πρώτος ε, διορθωτικός προπολογισμός. Ε, στις 5 Ιουνίου παρουσιάστηκε από τον κύριο Έτου τον Επίτροπο και παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας παρουσιάσει ο κύριος Ουρέλ. Ευχαριστώ. By Πρώτη φορά παίρνω το λόγο και θέλω να σας συγχαρώ εσάς και τους αντιπροέδρους για την επιτυχή σας εκλογή ορισμό την περασμένη εβδομάδα. Ε, σίγουρα μπορείτε να υπολογίζετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ε, έντιμη και εφοσιωμένη συνεργασία. Ε, ε, αυτό το εγχείρημα γίνεται κάθε χρόνο και αφορά ε, τη καταγραφή στον προπολογισμό των πλεονασμάτων ε, των περασμένων ετών. 15 Απριλίου κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται από το Δημοσιονομικό Κανονισμό, δηλαδή 15 μέρες μετά το κλείσιμο των λογαριασμών στις 31 Μαρτίου. Φέτος το πλεόνασμα είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2018, εκ των οποίων 1,3 δις προέρχονται από τα έσοδα του προϋπολογισμού, ενώ το μισό δις από τις δαπάνες. 1,3 δις από τα έσοδα προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από πρόστιμα ανταγωνισμού και άλλες κυρώσεις ε, και τόκους που ήδη ε, ε, πέρυσι. Όλα τα υπόλοιπα από τα έσοδα ε, αντισταθμίζουν το ένα το άλλο. Ας πούμε, οι τελωνιακοί δασμοί ε, ξεπέρασαν 160 εκατομμύρια το προβλογισμό. Απ' την άλλη είχαμε ενδεικτικό αντίκτυπο 200 εκατομμύρια λόγω ισοτιμιών. Από τις δαπάνες είχαμε υποεκτέλεση του προϋπολογισμού ε, σε όλα τα θεσμικά όργανα, πάνω από μισό δις σε ό,τι αφορά το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτελέστηκε στο 99,8% που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ε, εγγράφεται στο προϋπολογισμό λοιπόν το πλεόνασμα εφόσον εγκριθεί και αυτό θα σημάνει ότι θα μειωθούν οι συνεισφορές των κρατών μελών κατά το ίδιο ποσό, 1,8 δισεκατομμύρια. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Βιρέλ. Θα παρακαλούσα τον εισηγητή μας, τον κύριο Χάουερτ, να σχολιάσει αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν να ξεκινήσω σχολιάζοντα αυτή την ε, εισήγηση, θα ήθελα να προσθέσω τις ευχαριστίες μου και την εκτίμησή μου για την εργασία του προκατόχου μου, του Τανιέλε Βιώτη, ως ε, εισηγητή για το τμήμα 3 του Γενικού Προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019. Ο Ντανιέλε όχι μόνο διευκόλυνε την ε, ομαλή διαδικασία εδώ σε αυτήν την Επιτροπή, που θα έχετε εσείς φέτος Πρόεδρε την πρόκληση να αντιμετωπίσετε, αλλά ε, δείχθη ιδιαίτερα αποφασισμένος και αποτελεσματικός διαπραγματευτής ε, στις διαπραγματεύσεις, του σκαρπούς των οποίων θα δούμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης. Τώρα, τα θέματα αυτού του διορθωτικού προπολογισμού είναι διακριτικά θέματα που σημαίνουν κάποιες ε, τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια του ε, Στρασβούργου το Δεκέμβριο του 2018. Ε, επίσης, πρόκειται για θέματα τα οποία πρέπει να εκρίνουν ε, οι δημοσιονομικές αρχές. Ε, γι' αυτό και το συζητάμε σήμερα. Το πρώτο σχέδιο υποβλήθηκε τον Ιούνιο, στις 15 Ιουνίου, στην προηγούμενη θητεία και συνεχίζουμε σήμερα με την παρουσίαση σχεδίων εκθέσεων για αυτά τα τρία ε, σημεία και νομίζω η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 25 Ιουλίου και θα ψηφιστούν στην συνεδρίαση της Επιτροπής του Προϋπολογισμού στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου για να εγκριθούν μετά στην Ολομέλεια του ε, Σεπτεμβρίου. Είναι ένα τεχνικό θέμα, ε, ένα ακόμα 490 δις φτάνουμε στο 1,8 δις ε, όπως μας παρουσίασε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ωστόσο, εξής να σημειώσουμε πως είναι η θέση του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι παραμένει η ίδια μέχρι ότου αλλάξουμε ότι τα έσοδα από πρόστιμα κυρώσεις στον προπολογισμό δεν θα πρέπει απο, ε, απαραίτητο να οδηγήσουν στην μείωση των συμβολών των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να διατεθούν στον προπολογισμό. Και αυτή είναι η θέση μας. Στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτής η συμβολή θα πρέπει να αυξήσει με αντίστοιχο ποσό το αποθεματικό της Ένωσης όπως αυτό προτείνεται και να ε, απορροφηθούν όταν χρειαστεί. Επίσης υπάρχουν πρόστιμα σε, για υποθέσεις που είναι υπό εξέλιξη και διερωτώμε αν η Κομισιόν μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις για το τι περιμένει και ποιες είναι οι προσδοκίες όσον αφορά το πότε και το πόσο μπορεί να είναι αυτά τα πρόστιμα πράγμα που οποίο μπορεί να συμβάλλει στα έσοδα του προπολογισμού 2020, ώστε αυτό να αυξηθεί ε, σημαντικά. Αυτά έχω να πω και συστήνω να υποστηρίξουμε το πρώτο διευθυντικό προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, βουλευτές που θέλουν να σχολιάσουν αυτές τις δύο σύντομες εισηγήσει που ακούσαμε. Εφόσον όχι, Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να τονίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών έχει οριστεί στι 25 Ιουλίου στι 12 το μεσημέρι και ότι δεδομένε τη χρονική πίεση οι τροπολογίε αυτέ μπορούν να κατατεθούν μόνο στα αγγλικά. Mm. Ωραία λοιπόν, τότε να προχωρήσουμε στο σημείο 4 η διαδικασία. Θα ζητήσω στον κύριο Ρέλ της Επιτροπής να μας κάνει μια σύντομη ε, εισήγηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο κ. Χάουρτ, το σχέδιο διευθυντικού προπολογισμού 2 αποτελεί το follow-up της συμφωνίας του Δεκεμβρίου για τον προπολογισμό του 2019. Στη συμφωνία αυτή, τα θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν σε μια κοινή δήλωση να ενισχύσουν με 100 εκατομμύρια ευρώ τα προγράμματα Οριζόντας 2020 και το Erasmus+. Σε αυτή την κοινή διακήρυξη δεν δόθηκαν ενδείξει σε σχέση με την ε, κατανομή των 100 εκατομμυρίων μεταξύ των δύο προγραμμάτων και επομένω, η Κομισιόν θεώρησε ότι είναι λογικό να προτείνει μια ενίσχυση που να ακολουθεί το σχετικό μέγεθος των δύο προγραμμάτων, δηλαδή 80-20. Η πρόταση της Κομισιόν λαμβάνει επίσης ε, υπόψη την δυνατότητα απορρόφησης των προγραμμάτων αυτών. Τώρα, τα 80 εκατομμύρια της ε, ενίσχυσης που προτείνεται για τον ορίζοντα 2020 θα υποστηρίξουν ε, την έρευνα σχετικά με το κλίμα και πιο συγκεκριμένα τις ε, μεταφορές και τις μελλοντικές αναδυόμενες τεχνολογίες υπό το πιλωτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κοινοτομία. Σε ό,τι αφορά την έρευνα σχετικά με το κλίμα και τη σχετική πρόταση, η Κομισιόν λαμβάνει πρόφαση τι προτεραιότητε που εκφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολάκης. Με τον τρόπο αυτό, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού θα συνεισφέρει στο να ε, προσεγγίσουμε το συνολικό στόχο 20% για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής για την περίοδο 2014-2020. Ό,τι αφορά το Erasmus Plus, τα πρόσθετα 20 εκατομμύρια θα ενισχύσουν δραστηριότητες ε, στον τομέα του ΣΕ. Ανώτερης εκπαίδευσης, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ουρέλ. Κύριε Χάουαρτ. Ναι, πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού διαφέρει κάπως γιατί ε, παρόλο που είναι τεχνικό μέτρο, υλοποιεί την ε, Συμφωνία Συνδιαλλαγής για τον προπολογισμό του 2019. Και πράγματι συμφωνήθηκε ότι το Εράσμο και ορίζοντα 2020 θα ενισχυθούν με 100 εκατομμύρια συνολικά Αυτά θα ε, παρουσιάζονταν στην Δημοσιονομική Αρχή και αυτό γίνεται σήμερα. Επίση, συμφωνήθηκε σε συζητήσει εκείνε ότι αυτή η χρηματοδότηση θα αποτελούσε νέο χρήμα για αυτά τα νέα προγράμματα. Το σχέδιο του προπολογισμού 2 αντικατοπτρίζει την εκτέλεξη αυτή τη διευθέτηση. Ακούσατε την εξήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτή την διαίρεση των κονδυλίων. Ε, υπήρξε ε, μια συζήτηση, όχι πολύ συγκεκριμένη, αλλά ήταν καλό να γίνει αυτή η κατανομή βάσει του μεγέθους των προγραμμάτων, αλλά και της ικανότητας ε, να δαπανηθούν τα κονδύλια. Στην περίπτωση του ορίζοντα, 2020 τα ερευνητικά προγράμματα για το κλίμα τα κολοσορίζουμε. Εγώ ε, αναλαμβάνω δεσμευσή για το υπόλοιπο έτος. Ε, θα θυμάστε, όσοι ήσασταν εδώ στις 5 ε, Ιουνίου, θέσαμε κάποια ερωτήματα για την παρουσίαση του Επιτρόπου Έτιγκερ σε σχέση με το αν υπήρξε ε, ουσιαστικά κάποια παράληψη για τις ε, πιστώσεις πληρωμών. Δεν υπάρχουν πιστώσεις πληρωμών γιατί κυρίως στην περίπτωση του ορίζοντα, οι πληρωμές για τα προγράμματα αυτά θα προκύψουν τα μελλοντικά έτη. Και καθώς ε, θα προχωρούμε στον προϋπολογισμό, θα δείτε ότι αυτό είναι ένα μοντέλο για τα μεγαλύτερα προγράμματα. Και αναφέρεται λεπτομερώς στην έκθεση ότι τα κονδύλια για το Εράσμους μπορεί να ε, δοθούν νωρίτερα μέσα στο έτο και ίσω να θέλει να μα ε, δώσει εξηγήσει η Κομισιόν γιατί δεν έχουμε πιστώσει πληρωμών σε σχέση με το Εράσμους. Τι θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό στο μέλλον. Διαφορετικά θα έλεγα να υποστηρίξουμε αυτό το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού στα πλαίσια της ε, συμφωνίας ε, συνδιαλλαγής και την έγκριση του προπολογισμού για το 2019. Ευχαριστούμε κύριε Χάουαρτ. Υπάρχουν σχόλια για το σχέδιο αυτό. Υπάρχουν δύο. Και πάλι μπορώ να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ερώτηση που έθεσε μόλις ε, ο κύριος Χάουαρτ. Σε σχέση με τις πληρωμές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημείωσα την ερώτηση του εισηγητή και για τα πρόστιμα και τη μελλοντική τους εξέλιξη σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο του επιλογισμού θα σας δώσουμε πληροφορίες γραπτός για το θέμα αυτό. Τώρα, για αυτό το σχέδιο του διορθωτικού προπολογισμού. Όντω, τα 20 εκατομμύρια προ των κονδυλίων για το Εράσμους θα απαιτήσουν κάποιες πληρωμές φέτος, όμως είναι τόσο μικρό το ποσό και η Κομισιόν πιστεύει ότι κατά πάσα πιθανότητα μπορούμε να το καλύψουμε αυτό στο πλαίσιο του μελλοντικού εγχειρήματος ε, της επεγκόσμιας μεταφοράς ε, για τα νέα μέλη της Επιτροπής. Πρόκειται για ετήσια διαδικασία, προτείνει η Κομισιόν στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να μεταφέρει πιστώσεις πληρωμένων προγράμματα από όπου χρειάζονται λιγότερο και που χρειάζονται περισσότερο. Έτσι λοιπόν προτείνουμε να καλύψουμε τις πρόσθετες ε, ανάγκες για το Εράσμου στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ουρέλ. Σχόλια, ερωτήσεις, παρακαλώ, από τους βουλευτές. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 5. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα να κάνουμε μια κοινή συζήτηση για τα σημεία 5 και 6, γιατί συνδέονται στενά. Σε σχέση με το σημείο 5, λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μουρεσάν, τον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας επικοδομητικό χρόνο στην Επιτροπή Προλογισμού, όχι βέβαια κατά τη διάρκεια των διακοπών, μετά τις διακοπές τα επόμενα έτη. Τώρα, θέλω να αναφερθώ σε ένα απλό θέμα σήμερα το απόγευμα και προτείνει την ενεργοποίηση 293,6 εκατομμυρίων από το Ταμείο Αλληλεγγύης λόγω φυσικών καταστροφών στην Αυστρία, στη Ρουμανία και την Ιταλία που έλαβαν χώρα το 2018. Θα ήθελα να σας πω τι συνέβη ξεχωριστά στις τρεις χώρες γιατί χορηγούμε αυτά τα ποσά 8,19 εκατομμύρια ευρώ στη Ρουμανία για ζημιές από πλημμύρες στο δεύτερο ήμιση του έτους 2018. Συνολικές ζημίες ε, ήταν 327 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,7% του ΑΕΠ ε, της ε, βορειοανατολικής περιφέρειας της Ρουμανίας. Θα θυμάστε, συνάδελφοι, ότι προκειμένου το Ταμείο Αλληλεγγύης να μπορεί να ενεργοποιηθεί, να κινητοποιηθεί, πρέπει να πληρούνται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια. Είτε χρειάζεται να έχουμε μείζωνα φυσική καταστροφή σε ένα κράτο μέλο τη Ένωση, δηλαδή τουλάχιστον 0,6% του καθαρίστων χωρί εισοδήματο. Αυτή είναι μία, από είναι μία προποθέσει. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μία περιφερειακή φυσική καταστροφή που ισχύει αν τουλάχιστον 1,5% του ΕΕΠ της περιφέρειας ε, πλήττεται. Αυτό ισχύει για την αίτηση της Ρουμανίας και γι' αυτό εμπίπτει σε αυτή τη δεύτερη προϋπόθεση. Τρίτη προϋπόθεση, όταν κινητοποιούμε το Ταμείο Αλληλεγγύης, είναι αν για ένα ε, ε κράτος που συνορεύει σε μια χώρα που έχουμε μείζωνα φυσική καταστροφή. Αυτές είναι οι τρεις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του Ταμείου Λεγγύης. 327 εκατομμύρια ευρώ, ζημιά στη Ρουμανία, 2,7% του ΑΕΠ αυτής της περιοχής, οι πλημμύρες, καταστρέψαν υποδομές όπως ε, παραδείγματο χάρη, αναχώματα, φράγματα, ε, υποδομές ε, σε ό,τι αφορά το είδωρο και υποδομές σε ό,τι αφορά την γεωργία το 8,19 εκατομμύρια θα αποζημιώσουν δαπάνες για έκτακτη ανάγκη και για επιχειρήσεις ε, ανάκτησης και επίσης ε, για την προστασία της υποδομής και την αποκατάσταση της υποδομής για την Ιταλία. Προτείνουμε την κατανομή 277,2 εκατομμύρια ευρώ τι συνέβη στην Ιταλία. Επίσης είχαμε πλημμύρες, κατολιστήσεις και φυσικές καταστροφές που προκάλεσαν 34 θύματα το 2018 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικές ζημιές. Είχαμε δηλαδή μια μείζωνα φυσική καταστροφή εκεί. Τα 277 εκατομμύρια που εκταμιεύουμε θα χρησιμοποιηθούν για να ε, διασφαλίσουμε τις υποδομές ε, και θα δοθεί και ένα κονδύλιο. Ε, θα θυμάστε ότι με μέχρι 3 δισεκατομμύρια ζημιά μπορούμε να αποζημιώσουμε 2,5% της ζημιάς και 6% αν έχουμε πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Έτσι λοιπόν στην περίπτωση της εταιρείας έχουμε 2,5% και έχουμε 6% αν έχουμε 3 εκατομμύρια και πάνω. Δηλαδή 277 εκατομμύρια συνολικά. Τώρα για την Αυστρία Εκτεβιεύουμε 8,15 εκατομμύρια για καιρικά φαινόμενα κρέα που έλαβαν χώρα στη γειτονική χώρα. Η Αυστρία δεν εμπίπτει σε καμία από τις δύο κατηγορίες. Δεν ε, είχε φυσική καταστροφή, ούτε μίζωνα φυσική καταστροφή, όμως είναι όμορφη χώρα στην Ιταλία που χτυπήθηκε από μια μεγάλη φυσική καταστροφή και πληρούσε τις προποθέσει. Η συνολική ζημιά ήταν 326 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα που εκταμιεύουμε ε, έχουν ε, να κάνουν με μέτρα για να αποφύγουμε τη διάβρεση του εδάφους, αλλά και να έχουμε και επιχώματα σε ποτάμια, να έχουμε σε ποτάμια. Αυτό αφορά το πεδίο εφαρμογής των εκταμιεύσεων να πω συνάδελφα ότι και τα τρία κράτη-μέλη έχουν υποβάλει εγκαίρως τις αιτήσει 12 εβδομάδες μετά τις φυσικές καταστροφές μέσα σε 12 εβδομάδες αυτό ισχύει 7 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα της Ρουμανίας 20 Δεκεμβρίου και η Ιταλία και 14 Ιανουαρίου η Αυστρία αξιολόγησε η Κομισιόν τις αιτήσει και όλες συνάδουν με τις απαιτήσει και γι' αυτό η Κομισιόν προτείνει και υποστηρίζει να εκταμείευσουμε αυτά τα ποσά κατά προτεραιότητα. Και γι' αυτό, Πρόεδρε, προτείνω να δράσουμε γρήγορα. Καλούνται οι συνάδελφοι να καταθέσουν τροπολογίες μέχρι τις 25 Ιουλίου, την 5η δηλαδή, προς το τέλος της εβδομάδας. Και η ψηφοφορία προβλέπεται στις 3 Σεπτεμβρίου και κατόπιν στην Ολομέλεια στη, του Σεπτεμβρίου, που είναι η πρώτη ολομέλεια που θα έχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μουρεσάν κύριε Χάουαρτ. Δεν θα σας εκπλήξει ότι και εγώ συνιστώ να υποστηρίξουμε το διορθωτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό να κινητοποιηθούν τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Αλληλεγγύης για να αντιμετωπιστούν αυτές τις συμφορές και τα δεινά που μας είπε ο κύριος Μουρεσάν. Τον ικανοποιεί και τον ίδιο η πρόταση αυτή, υποθέτω, και ε, σα συστήνω να εγκρίνουμε αυτή τη δαπάνη. Σε σχέση με αυτό το διορθωτικό προπολογισμό συμφωνεί και το Συμβούλιο και προτίθεται στις 3 Σεπτεμβρίου να εγκρίνει με την ταχεία διαδικασία αυτό το ποσό. Ευχαριστώ κύριε Χάουαρτ. Θέλει κανείς να σχολιάσει, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα. Θέλουμε να συγχαρούμε τον εισηγητή για το έργο του για το θέμα αυτό. Υποστηρίζουμε την πρότασή του. Απλώς ήθελα να σας πω ότι είμαι μέλος της Επιτροπής, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και του προπολογισμού και πιστεύω ότι πλέον οι έκτακτες καταστάσεις δεν είναι έκτακτες, είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και σε σχέση ε, με το ε, δημοσιονομικές προοπτικές, το PDP, ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό το ταμείο, και το ταμείο αλληλεγγύης, αλλά και της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε έτσι πιο μακροπρόθεσμα και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μάλιστα, όλοι σας άκουσαν, ήσασταν σαφέστατος και ξεκάθαρος, παρακαλώ. Ναι, και εγώ θέλω να σας καλωσορίσω όλους και εγώ υποστηρίζω τον εισηγητή μου Ρεσάν. Η κατάσταση είναι αυτή που μας θύμισε. Πραγματικά ήταν δραματικές οι συνθήκες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μου όλος ιδιαιτέρως ε, υπέφεραν διάφορες περιφέρειες, κυρίως η Βόρειο-Ανατολική, με φοβερές ε, ε, καταστροφές. Ε, που κατέστρεψαν πάνω από 400.000 εκτάρια ε, ε, Natura 2000, δηλαδή ευαίσθητα οικοσυστήματα. Ευχαριστώ και ελπίζω να πάνε τα πράγματα γρήγορα. Okay, thank you. Any more comments? If... Άλλα σχόλια παρακαλώ. Όχι. Ωραία, τότε το 5 και το 6 τα κλείσαμε. Να τονίσω ωστόσο ότι το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 3 ακολουθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα όπως το 2 και το, 1, δηλαδή ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας το 3 Σεπτεμβρίου. Πάμε στο σημείο 4. Αντίθετα με τα προηγούμενα, ε, σημείο 7, ε, έχουμε το διορθωτικό προπολογισμό 4 που εγκρίθηκε στις 2 Ιουλίου από την Επιτροπή και ε, όμως δεν είχε παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Ρίλ να μας κάνει μια σύντομη εισήγηση ε, σε σχέση με αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ, ευχαρίστως. Διορθωτικός προϋπολογισμός ε, νούμερο 4. Εισάγει διάφορες τεχνικές ε, προσαρμογές και από την πλευρά των εσόδων και από την πλευρά των δαπανών του προϋπολογισμού ε, κατόπιν της οριστικοποίησης κάποιας νομοθετικής διαδικασίας και χάρη στην αξιολόγηση των αναγκών μέχρι το τέλος του έτους καθώς και ενημέρωση των προβλέψεων σε σχέση με τους ίδιους πόρους και σχετικές διορθώσεις. Θα δείτε εδώ στο σχέδιο δοτικού προπολογισμού τρία βασικά συστατικά. Το πρώτο αφορά το τμήμα του προπολογισμού για την Κομισιόν στο κομμάτι των δαπανών που προτείνουμε διάφορες ε, προσαρμογές. Οι πιο σημαντικές είναι οι εξής μείωση 18,5 εκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Εποπτική, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές μετά από την ολοκλήρωση της αναθεώρησης των εντολών τους. Όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έφτασαν σε συμφωνία για την αναθεώρηση αυτών των εντολών, κατέστησε σαφές ότι οι δημοσιονομικοί φάκελοι που αρχικά είχαν προβλεφθεί από την Κομισιόν για αυτή την αναθεώρηση ήταν μεγαλύτερη και άρα λοιπόν η μείωση 18,5 όπως σας είπα αντικατοπτρίζει την μείωση της τελικής αναθεώρησης των εντολών. Δεύτερον, περίπου 19 εκατομμύρια είχαν μείνει στο αποθεματικό για την ε, οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex ε, συνοριοφυλακή και ακροφυλακή λόγω του ότι η νέα βάση για αυτόν τον οργανισμό του Frontex και πιο συγκεκριμένα η πρόσληψη των ε, περίφημων 10.000 συνοριοφυλάκων για τους οποίους ε, θα αρχίσει να ισχύει η νομική βάση αργότερα από ό,τι αναμενόταν ε, αυτό μας επιτρέψει να απελευθερώσουμε ή μάλλον να ακυρώσουμε 12,2 εκατομμύρια από αυτό το αποθηματικό. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν συστατικό. Το τρίτο συστατικό αφορά ένα διαφορετικό αποθεματικό 460 εκατομμύρια είχαν μπει στο αποθεματικό στον προπολογισμό του 2019 για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου από αυτό το ποσό ένα πρώτο κομμάτι 370 εκατομμυρίων είχε δει απολευθερωθεί μέσω μιας μεταφοράς το Μάρτιο. Μια δεύτερη δόση 32,8 εκατομμυρίων προτείνεται αυτή τη στιγμή από την Κομισιόν για απελευθέρωση και αυτό το έχετε ενώπιόν σας. Θα ψηφίσετε γι' αυτό αύριο και έτσι έχουμε ένα μικρό ποσό 7,2 εκατομμύρια που μένουν στο αποθεματικό και τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν επίσης να ακυρωθούν γιατί πιστεύουμε ότι με τα τρία ποσά, τα 370 και τα 82,8 μπορούν να καλυφθούν παρκώς ε, οι ανάγκες. Έχουμε και το αποθηματικό για το REST EU. Μια συμφωνία επί της νομικής βάσης επετέφθη μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου περί τα τέλη του περασμένου έτους και το ποσό επί το οποίο έγινε η συμφωνία ήταν χαμηλότερο από αυτό που αρχικά πρότεινε η Κομισιόν. Άρα λοιπόν και αυτό αν θέλετε είναι μια λογική συνέχεια της συμφωνίας ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και την μείωση του 2019 που αφορά 35 εκατομμύρια. Τελευταία σημαντική συνιστόσα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης όπου ένα ποσό του ύψους των 29,7 εκατομμυρίων είναι διαθέσιμο για προκαταβολές και αυτόματα μεταφέρθηκε από το 2018 στο 2019 μετά από μια νέα διάταξη στο αναθεωρημένο, στον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό εφόσον ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει ότι το σύνολο ποσό για προκαταβολές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια. Με αυτόν τον διορθωτικό προπολογισμό προτείνουμε την μείωση κατά 29,7 εκατομμύρια και άρα να επανέλθουν στα 50 εκατομμύρια οι ε, διαθέσιμες πιστώσεις. Επόμενο συστατικό αφορά προσαρμογές που αφορούν άλλους θεσμούς και ακολουθεί την αναβολή της ε, εξόδου του Ευρωπαϊκού Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν υιοθετήθηκε ο προπολογισμό του 2019, είχαμε θεωρήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποσυρώταν από, το, από την Ένωση στα τέλη Μαρτίου και αυτό θα σήμαινε οικονομικές επιπτώσεις για διάφορους θεσμού. Όμω τώρα που η αναβολή θα πάει μάλλον, μάλλον είναι γεγονός μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, αυτοί οι θεσμοί τώρα ζητούν να αντιστραφούν αυτές οι αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά αύξηση 15,1 εκατομμύρια στον προπολογισμό του. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά 0,1 εκατομμύρια. Και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, της οποίας ο προπολογισμός είχε αυξηθεί εν ώψη εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου το Μάρτιο, τώρα επιστρέφει κάποια ε, περιτά χρήματα, ε, δηλαδή 3,3 εκατομμύρια. Για να κλείσουμε λοιπόν τώρα, έχουμε τα έσοδα του προϋπολογισμού Στην άλλη πλευρά, ενημέρωση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του 2019 μετά από τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για τα δεδομένα GNI και ε, ΑΕΠ και ΦΠΑ προβλέψεις δηλαδή για τη συλλογή των ε, δασμών ε, αυτών. Ε, η Συμβουλευτική Επιτροπή Περιπόρων συναντήθηκε στις 25 Πέμπτου του τρέχοντος. Τώρα, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τακτικά και έτσι οι συμβολές των 100 μελών ε, είναι πιο σύμμορφες με τα ποσά που τελικά θα οφείλουν. Ως αποτέλεσμα αυτής της ετήσιας ενημέρωσης, οι εξπόστ δημοσιονομικές προσαρμογές είναι εν γέννη μικρότερες. Αυτά είχα να πω και έτσι τελειώνει η εισήγησή μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ιουρέλ. Ο κύριος Χάουαρτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ιουρέλ για την παρουσίασή του των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού είναι ελαφρώς, μάλλον αρκετά διαφορετικό από τα τρία προηγούμενα που μας απασχόλησαν. Πρώτον, είναι πολύ πιο περίπλοκο από τη φύση του, καλύπτει ε, πολλές θέσεις του προϋπολογισμού, αλλά το πιο κρίσιμο είναι ότι μόλις σήμερα λάβαμε αυτά τα στοιχεία, ενώ εγώ μόλις την περασμένη εβδομάδα ορίστηκα διάδοχος ε, και του κυρίου Βιώτη. Οπότε δεν είμαστε σε θέση να το μελετήσουμε επαρκώς. Το χρονοδιάγραμμα που προτείνω. Bring the Να ε, υποβληθεί η προσυζήτηση στην Επιτροπή Προπολογισμών στις 2 ή 3 Σεπτεμβρίου με τις τροπολογίες να κατατίθενται προς τα τέλη εκείνης της εβδομάδας και να ψηφιστούν τέλη Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα επειδή η πρόταση αυτή, όπως σας είπα, είναι αρκετά περίπλοκη. Πολλά μέλη της Επιτροπής μας είναι νέα και θα ήθελα να έχουν χρόνο να τα μελετήσουν. Τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα είναι μάλλον τεχνικά και δεν υπάρχουν ζητήματα ε, εκροών και εκταμιεύσεων για ε, τα θεσμικά όργανα. Το Συμβούλιο μπορεί να ακολουθήσει στις 6 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπετε, ε, τη διαδικασία και να το εγκρίνει, αλλά δεν θα ήταν σωστό σε αφορά το δικό μας λόγο, δηλαδή να παρακάμψει την κανονική διαδικασία, γιατί είμαστε και εμεί σκέλο τη Δημοσιονομική Αρχή. είναι Ολομέλεια θα συζητηθούν αυτά τέλη Οκτωβρίου. Υπάρχει χρόνο να τα εξετάσουμε και να τα συζητήσουμε ενδελεχώ. Ευχαριστώ. Σχόλια, ερωτήσει, παρατηρήσει. Ε, κλείνω λέγοντα αυτά που είπε και ο εισηγητή, ότι θα καταθέσει σχέδιο εκθέση στι 2 3 του Σεπτέμβρη ε, και να ψηφίσουμε ε, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ε, ε, ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 8. Πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κινητοποίηση ε, κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση για τεχνική αρρωγή. θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Ράνζα, για να μα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου, ε, η έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ε, η αγορά εργασίας ε, αλλάζει υφίστανται συνέπειες και επιπτώσεις ε, οι εργαζόμενοι και οι αυτοπασχολούμενοι και όλοι οι φορείς ε, της αγοράς εργασίας. Έχουμε διάφορες διαδικασίες ανασυγκρότησης ε, όπου οι εργαζόμενοι απολύονται. Έχουμε λοιπόν αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να βοηθάει τους εργαζομένους να μπορούν να εντάσσονται ξανά στην αγορά εργασίας. 150 εκατομμύρια ευρώ είναι ε, η οροφή ε, από το 2011 ε, από τότε που δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο ταμείο έχει αλλάξει πολλές φορές ο τρόπος που εφαρμόζεται. Σήμερα είμαστε στο 60% σύμφωνα με τον αντίστοιχο κανονισμό μπορεί να δοθεί ως τεχνική βοήθεια ετησίως μόνο μισό της εκατό. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, με ε, την πρόταση και το αίτημα 600.000 ευρώ για το 2019. Πρόκειται για τεχνικές δαπάνες. Ε, προς ποια κατεύθυνση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόκειται πρώτα απ' όλα για συλλογή στοιχείων και δεδομένων, τα οποία χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί ε, και ε, στα οποία έχει δοθεί συνέθεια με κάποια κονδύλια που ε, εκταμιεύτηκαν και τα συγκεκριμένα μέτρα. Για να συλλεγούν λοιπόν αυτά τα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αφιερώσει 20.000 ευρώ. Δεύτερον, υπάρχει στο σελίδα, ε, στο τοπό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που θα πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πάλι 20.000 ευρώ είναι το κόστος εκεί. Το προβλεπόμενο κονδύλι, ε, ε, αυτό ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτο μέτρο βελτίωση ανταλλαγής δεδομένων και των αντιστοίχων συστημάτων και μείωση των χρόνων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υποβολή αιτημάτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το σκοπό αυτό έχει προβλέψει για την ανταλλαγή των δεδομένων 80.000 ευρώ. Επίσης, ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 70.000 ευρώ να ε, δοθούν για ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα συνεδριάσουν δύο φορές το 2019 και μετά ε, στο πρώτο εξάμεινο το 2020. Ποιοι είναι αυτοί οι εμπειρογνώμονε, πρόσωπα από, διάφορα, από όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από κάθε κράτο. Και επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα κονδύλι 70.000 ευρώ άλλο που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τεχνική υποστήριξη και διοικητική υποστήριξη, θέλει να διοργανώσει δύο σεμινάρια για τους κοινωνικούς εταίρους, τα οποία κοστίζουν 120.000 ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Πρόκειται για σεμινάρια για τη δημιουργία δικτύου επαφών. Αυτά. Ε, και θα είναι τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει κάτι ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται για την εκ των αξιολόγηση, έχει εκ των προτέρων και έχει προβλέψει 300.000 0,35% είναι το ποσό του ετήσιου προπολογισμού, 610 εκατομμύρια. Δεν ξεπερνάμε χιλιάδες, συγγνώμη, 610.000. 610.000. Δεν ξεπερνάμε το πλαφόν. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται επικρίσεις για αυτή την ε, υπέρογγη διοικητική μηχανή. Το Ταμείο αυτό όμως λειτουργεί και θέλουμε να λειτουργεί ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο αποτελεσματικά. Και θεωρούμε ότι τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξίζει να υποστηριχθούν. Και θα πιάσουν και τόπο, είμαι βέβαιος, στα χρήματα αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά προσωπικά σας συνιστώ να εγκρίνουμε ε, αυτή τη δαπάνη. Ελπίζω να μην πέρασα και το πεντάλεπτο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε τον κύριο Σιγητή. Υπάρχουν σχολεία ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά για την παρουσίαση αυτή. Μια ερώτηση σε σχέση με τη συνεδριάση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων. Αναφέρεται εκεί το ποσό των 70.000 ευρώ. Μπορούμε να ξέρουμε πόσες μέρες συνεδριάζουν οι εμπειρογνώμονες ε, και την τοποθεσία των συνεδριάσεων ε, και πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων πράγματι θα χρησιμοποιηθούν ε, με το βελτιστό δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να λάβουμε απάντηση σχετικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Przedstawiciel Komisji udzielił tej να δώσουμε το λόγο πρώτα στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να απαντήσει. Παρακαλώ, κύριε Ουρέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, δεν ε, δίναμε να απαντήσω αμέσω ε, σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Θα σας στείλουμε μια γραπτή απάντηση σε σχέση με τον αριθμό και τις σχετικές λεπτομέρειες των συνεδριάσεων Ομάδας επιρρογνωμόνων. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Άλλες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Επομένω πάμε στο σημείο 17. Θυμάστε ότι έχουμε κάνει μια τροποποίηση, μια αλλαγή στην αρχή της συνεδρίασης και ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας. Εισαγωγικά Καταρχήν, ε, να σας πω ότι μία σειρά σημειωμάτων ε, για το ιστορικό έχουν κυκλοφορήσει από την Κομιτεία σχέση με τους κύριους φακέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού και παρουσιάζουν την κατάσταση σε διάφορους φακέλους. Θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια και κατόπιν κάποια περαιτέρω σχόλια. Καταρχήν, ε, ε, οι βασικές ε, και επαναλαμβάνομες εργασίες αυτής της Επιτροπής είναι φυσικά η ετήσια δικασία χαράξη του προπολογισμού που αποτελείται από τρεις ή τέσσερις ε, κύκλους, τα σχέδια προπολογισμών, τους προπολογισμού που υφίζονται και τους εκτελεσμένους προπολογισμού. Επίσης, θα ασχοληθούμε με στρατηγικά νομοθετήματα που συχνά συσχετίζονται σε συνεργασία με άλλες επιτροπές, πριν την εφαρμογή του ΕΦΣΙ, του InvestEU, το πρόγραμμα υποστήριξης μεταρρυθμίσεων ή άλλες πρωτοβουλίες για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Τρίτη. Παρατήρηση έχει να κάνει με το Brexit ε, που μάλλον θα μας ε, κρατήσει απασχολισμένους ε, Έχουμε αντικτύπο, σε θέματα που αφορούν ε, τα κτίρια ε, και τους οργανισμούς ε, μέχρι και τη διαχείριση που θα υπάρχει αν υπάρχει απόσυρση με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία. Στην τελευταία περίπτωση θα χρειαστούν μέτρα εκτεκτής ανάγκης σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους, η βασική προτεραιότητα της επόμενου μήνε θα είναι όταν το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο ή η τελική συμφωνία για το πλαίσιο 2021-2027 θα συζητείτε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Είναι σημαντικό και επίγον να επανακινήσουμε τη δράση μας στο φάκελο αυτό. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Πάρα πολλή δουλειά έχει γίνει στην προηγούμενη θητεία για να πετύχουμε την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θετήθηκε στην Ολομέλεια του 2018, του Νοεμβρίου του 2018, με την ενδιάμεση έκθεση. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτές τις εργασίες για να διασφαλίσουμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο σημερινό σύστημα, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων ένα συνολικό ε, μέγεθο πολιτή δημοσιονομικού πλησίου στα 1,3 του ακαθαρίστου ε, εγχωρίου εισοδήματο με, διασφαλισμένου πόρου ε, και για καινούριε αλλά και πιο παραδοσιακέ πολιτικέ. Δεύτερον, ε, ενισχυμένε δυνατότητε ευελιξία και υποχρεωτική αναθεώρηση ενδιάμεση για να έχουμε περισσότερο περιθώριο λιγμών και να αντιμετωπίσουμε τις προτεραιότητες και τα πρόβλεπτα που μπορεί να προκύψουν σε αυτή την επιτετία. Και τέλος, νέους πόρους. Ακροπρόθεσμη προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν σχεδιαστεί καλά η μεταρρύθμιση των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ξεκλειδώσει τη μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά τις δαπάνες και να φέρει ωφέλη και για τι πολιτικέ και ξεκάθαρη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Οι θέσει ε, στο φάκελο του πολιτικού του δημοσιονομικού πλασίου βρίσκονται στο επίκεντρο τη ε, ε, νομοθετικής, διαδικαστική πολιτικού, διαδικαστικού, πολιτικού αγώνα εξουσίας για να είμαστε επιτυχείς χρειαζόμαστε συντονισμένη δράση εντός του Κοινοβουλίου με τις τομέικες επιτροπές, τη διάσκεψη των Πρόεδρων και φυσικά με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Επίσης θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τον διοργανικό διάλογο με το Συμβούλιο και να ξεκινήσουμε πραγματικές διαπραγματεύσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σέβονται την διαπραγματευτική μας θέση και να λαμβάνουν υπόψη τη συνεισφορά μας στην τελική συμφωνία αν είναι να πετύχουμε συνένεση. Βασίζομαι πολύ στην Προεδρία της Φιλανδίας και στην Κομισιόν ως διαμεσολαβητή για να διασφαλίσει ότι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σαφήνεια διαβιβάζονται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Και το πρώτο μήνυμα που θέλω να διαβάσω σήμερα είναι το εξή. Μια συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν είναι το τελικό βήμα στη διαδικασία. Η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι κάτι το τυπικό το κερασάκι σε όπως ε, το αποκαλούμε, θα πρέπει ε, να συνοδεύεται από ουσιαστική πρόοδο σε τομείς που είναι δικέ μας δικές μας προτεραιότητες. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία και μπορείτε να βασιστείτε σε μένα ως πρόεδρο της Επιτροπής αυτής ότι αυτό θα το ξεκαθαρίσω και θα υπονθυμίζω σε όλους τη θέση αυτή. Αυτή ήταν ε, η σύντομη εισαγωγή μου. Ίσως να ήταν κάπως μακροσκελής, ε, ίσως όχι για κάποιους. Θα ήθελα να ζητήσω τα σχόλιά σας για τα θέματα αυτά και φυσικά να ξεκινήσουμε από τους συντονιστές ε, και τους αρμόδιους συνταξεκθέσεων. Ποιος θέλει να σχολιάσει εγώ ως και συντονιστής αλλά και πρώην συνεισηγητής για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα να σχολιάσω τη δήλωσή σας, ξεκινώντας από το τελευταίο σημείο. Γιατί κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη, κυρίως εντός της Επιτροπής μας, ότι δεν ε, είναι μονόδρομοι οι επιλογές, δεν είναι ότι ε, θα πρέπει να δώσουμε τη συνένεση, θα δώσουμε την ε, συμφωνή γνώμη μας αν εγκρίνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και για το Συμβούλιο, γιατί Φυσικά το Συμβούλιο εργάζεται συνεχώς και δίωση η Φιλανδική Προεδρία και πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή θα προετοιμαστεί κοινή θέση για να διαπραγματευτούν κάτι που εμπίπτει στη δική μας αρμοδιότητα στο διαπραγματευτικό πεδίο κατόπιν. Θα έχουν τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που σχεδιστεί για το Δεκέμβριο και του χρόνου θα έχουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου που θα στελεί στο Κοινοβούλιο. Αυτέ οι δράσει υλοποιούνται και η δική μα προσέγγιση μέχρι τώρα ήταν να μην είμαστε παθητικοί. Γιατί σύμφωνα με τη συνθήκη θα πρέπει να περιμένουμε ε, το Συμβούλιο. Όμως ε, είμαστε ενεργητικοί. Για εμάς είναι σημαντικό να αναλάβουμε δράση αμέσως ε, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και να ενημερώσουμε το Συμβούλιο ότι αν δεν διαβουλευτούν με το Κοινοβούλιο, είναι πιθανόν, πάρα πολύ πιθανόν, ότι εμείς δεν θα συνενέσουμε, αν δεν υπάρχει δηλαδή σχετική διαβούλευση. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ευαισθητοποίηση για όλους τους συμμετέχοντες. Γιατί διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι το εξή. Θα μα φέρουν την κοινή θέση και θα μα πούν: Ακούστε, 27 πρωθυπουργοί κτλ. κτλ συμφώνησαν. Πώ μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι καλύτερα να τους ενημερώσουμε ότι από την αρχή θέλουμε ένα εργό ρόλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το συμπερασμά σας. Ένα πράγμα είναι η μεθοδολογία, αλλά και η προοπτική είναι σημαντική. Και είναι σημαντική γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο τέλος του 2020 και όχι στις αρχές του 2020. Το σχέδιο μας ήταν να είμαστε έτοιμοι πριν τις εκλογές. Ε, λοιπόν, ε, δεν είναι από τι εκλογέ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη την ισχύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επηρεάσουμε τη διαδικασία. Thank you very much. Madame Ευχαριστώ, Γουάρδια Σάμπαλ. Παρακολουθώντα αυτά που σχολιάσατε εσεί, για αυτά που είπε και ο κύριο Όλμπριχτ, είναι αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο έχει την ε, ε, εξουσία, αλλά όχι την υποχρέωση να συνέσει επί του πολίτη του μεσονομικού πλαισίου. Και ήδη ε, είχαμε ξεκινήσει και στην προηγούμενη διαδικασία. Πάντα λέγαμε στο Συμβούλιο ότι είναι, και λέγαμε ότι είναι πολύ πολύπλοκε οι εσωτερικέ διαπραγματεύσει. Αλλά όταν υπάρχει σε συμφωνία, πρέπει να έρθουν να διαπραγματευτούν με το Κοινοβούλιο και να πετύχουν αυτή την συνένεση του Κοινοβουλίου και αυτό ισχύει για οποιοδήποτε έργο της Επιτροπής Προπολογισμών και σε ό,τι αφορά και τον ετήσιο προπολογισμό. Γιατί όταν μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη νομοθετική έκθεση, η συναπόφαση λειτουργεί πολύ καλά, γνωμοδοτεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ολοποιεί τη δική του πρόταση και κάθονται στο τραπέζι και τα διόργανα να διαπραγματευτούν. Κάτι με τον προπολογισμό δεν συμβαίνει συνήθως και σχεδόν υπάρχει μια διαδικασία περισσότερο συνένεση παρά πραγματικής νομοθετικής διαπραγμάτευσης. Δεν είναι συναπόφαση, είναι συνδιαλλαγή. Όμως ε, τελικά μόνο ένα μέρος ε, της οικογένειας ε, συνδιαλέγεται και τελικά πάντα το Κοινοβούλιο πρέπει να υποχωρήσει για να υπάρξει συμφωνία. Αυτό είναι κάτι που το θέτουμε επιτάπητο συχνά, όμως τελικά ποτέ δεν ε, καταφέρνουμε ε, να διαβιβάσουμε το μήνυμα στο Συμβούλιο. Εγώ νομίζω ότι μία από τις πρώτες προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας όχι από τη σκοπιά των πολιτικών θεμάτων, αλλά για το πώς θα κάνουμε σεβαστή τη θέση του Κοινοβουλίου, είναι ακριβώς ότι θα πρέπει να μας δουν ως την άλλη δημοσιονομική αρχή. Είμαστε δύο που πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι και που θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να φτάσουμε σε συμφωνία αυτό ως ε, τρόπο εργασίας. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα. Προφανώς το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι προτεραιότητα, είναι επιτάπητος και οι αιτήσεις υπηρεπολογισμοί επίσης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τα επόμενα πέντε χρόνια. Ίσως να συμβούν πράγματα εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση που να μας θέσουν νέε προτεραιότητε επιτάπητο, όπως έγινε στην προηγούμενη θητεία. Όμω, ό,τι και να συμβεί, εγώ νομίζω τα θέματα τη κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση και των προσφύγων, η στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, θα είναι ούτω ή άλλω επιτάπητο. Και το ακούσαμε και τι προάλλε στην παρέμβαση της Ουρσουλα Φόντε Λάιεν. Ε, είπαν ότι αυτά θα είναι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι και προτεραιότητες αυτού του Κοινοβουλίου και από αυτόν θα πρέπει να συζητήσουμε. Και σε σχέση με όλα αυτά θα πρέπει να συζητήσουμε και πάρα πολύ για τη δική μας συνεργασία και την ανάπτυξη με την Αφρική, για το τι θα συμβεί με όλα αυτά τα νέα μέσα που θα συζητήσουμε και αύριο με τους οργανισμούς για το συνεργειακό έλεγχο και για το νέο σώμα των συνεργοφυλάκων. Γιατί ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί και στη συνέχεια τις ε, προτεραιότητες ε, που θα προκύψουν ε, τα επόμενα πέντε χρόνια ως έκτακτες. Νομίζω ότι σε αυτές τις γραμμές πρέπει να εργαστούμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Αντρέσεν. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. I want to add uh, Θα ήθελα να προσθέσω μερικά πράγματα από την προοπτική των πρασίνων. Έχει σημαντικό ρόλο η Επιτροπή μας και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να είναι ισχυρός ο προϋπολογισμός ε, και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τα θέματα που μας απασχολούν με το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Μπορεί να διαφέρουμε λίγο από τις άλλες επιτροπές, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι υπέρ ενό φιλοευρωπαϊκού ισχυρού προπολογισμού στι μάχε που έχουμε να δώσουμε με το Συμβούλιο. Το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με το μέγεθο του προπολογισμού, αλλά και με την ποιότητα του προπολογισμού. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν έχουμε πράξει, έτσι ώστε η Συμφωνία των Παρισιών ε, των Παρισίων και οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη να ενταχθούν στις διαπραγματεύσεις που έχουμε για τον προϋπολογισμό και τις αιτήσεις ενώ όλα και για το PDP. Ακούσαμε την κυρία Φόντρα Λάιεν την περασμένη εβδομάδα. Μίλησε για μια νέα πράσινη συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ως ύψιστη προτεραιότητά της την ανέφερε για τους επόμενους μήνες. Αυτό θα πρέπει να σημαίνει κάτι και για μας τη συζήτηση που θα κάνουμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά μπορεί να συνδεθεί και όλα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα άλλα θέματα που θα μας απασχολήσουν στην Επιτροπή μας. Και αυτό μου έλειψε λίγο από τα αρχικά σας λόγια κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτά τα θέματα που συνδέονται με το κλίμα ε, και τον προϋπολογισμό σημαίνουν πολλά για μας, τους πρασίνους και σου λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι προτεραιότητά της ε, των 100 πρώτων ημερών, άρα και εμείς θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Κυρία Αγίε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όλοι νομίζω συμφωνούμε για αυτά τα θέματα, συγκλίνουν οι απόψει μα. Θα ήθελα να θυμίσω, όπω οι συνάδελφοι προηγουμένω, ότι χρειάζεται το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο να είναι φιλόδοξο και ε, για να διατηρήσουμε ιστορικά τα κονδύλια της ε, ΚΑΠ και του Ταμείου Συνοχής απαντώντας όμως ταυτόχρονα και στις μεγάλες προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη πενταετία. Ξέρουμε ποιο είναι το πλαίσιο, ξέρουμε ποιες είναι οι προκλήσεις, έχουμε και το Brexit μπροστά μας ε, που τους επόμενους μήνες θα λυθεί κανονικά. Ε, μας καλούν όλους όλα αυτά για ένα φιλόδοξο PDP και συνδέεται με αυτό άμεσα, υπόθηκε προηγουμένως ότι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο συνδέονται με τους ίδιους πόρους. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον ε, ε, οι πολλοί νέοι εκλογέντες, εγγραφόμαστε σε αυτή τη ε, γραμμή για επιπλέον ιδίους πόρους. Είναι πολύ καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια βάση, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και παραπέρα ένα φόρο για το διοξίδιο του άνθρακα στα σύνορα ή φόρο ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Είναι ακόμα πολύ διστακτικό το Συμβούλιο. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη πυγμή και φιλοδοξία και χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Merci, Madame Mr.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 θα ήθελαν ε, η Επιτροπή μας να εγκρίνει ένα δραστήριο πρόγραμμα. Ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμα της ε, Επιτροπής, αλλά η Επιτροπή του Προπολογισμού είναι, μία από τις, είναι τις πιο σημαντικές. Όλες είναι σημαντικές, αλλά τα μάτια όλων είναι στραμμένα προς εμάς και στις χώρες μας. Εμείς πρέπει να εξηγήσουμε τι κάναμε, τι ιδέες ε, προτείναμε, ποιες ιδέες προέκυψαν από εδώ. Οπότε θα στηρίξω τις δραστηριότητε της Επιτροπής μας και κυρίως τον πρόεδρό μας που θα μας εκπροσωπήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε τις δικές μας λύσεις. Η Φιλανδική Προεδρία φαίνεται να ορίζει φιλόδοξους στόχους. Μιλάμε για νούμερα και ποσοστώσεις μετά τις διακοπές. πρέπει να προετοιμαστούμε. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει να μην υπάρξουν περικοπές στην πολιτική συνοχή, στη γεωργική πολιτική. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία, με την μετανάστευση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, να ας προετοιμαστούμε. Εγώ θα στηρίξω αυτό το είδος δραστηριότητας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Howard. Thank you uh, again. Ο κύριος Χάουαρτ. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα τη ιεράρχηση και των προτεραιοτήτων προπολογισμών θα ήθελα να τονίσω τρία-τριάμιση σημεία σε αυτό το πλαίσιο. Ε, τρία εκ των οποίων νομίζω θα απαιτήσουν ε, την στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού αυτής εδώ της Επιτροπής και πιστεύω ότι θα είναι και αυτονόητο γιατί η κλιματική δράση δικαίω και σαφώς θα είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον προπολογισμό της. Αλλά όπως δείχνουν, έδειξαν μάλλον οι ακροάσεις στην προηγούμενη θητεία, εάν δεν προσέξουμε αν όντως επιτυχάνουμε τους στόχους και ότι αυτοί οι στόχοι αποδίδουν με αλλαγές που εμείς θέλαμε να δούμε, τότε η εναλλακτική είναι τελικά τι να κάνουμε, να βάψουμε τα πάντα πράσινα. Δεν ενδιαφέρει όμως κανέναν ε, κάτι τέτοιο, όποια και είναι η πολιτική του πεποίθηση. Απλά δηλαδή να βάψουμε από πάνω με πράσινο χρώμα ό,τι κάνουμε. Θέλουμε τα χρήματα που δαπανούμε να έχουν και αποτέλεσμα, ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε μαζί με την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, ώστε να έχουμε σωστό δημοσιονομικό έλεγχο. Να βλέπουμε πώ δαπανώνται αυτά τα χρήματα. Τώρα, όσον αφορά τη συνοχή και το κλίμα, είναι σωστό το ότι συνδέαμε αυτά τα δύο πράγματα. Η συνοχή ανέκαθεν ναι, ήταν ένα μέσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να θέτει σε εφαρμογή τα ιδανικά τη. Σε πράξη, μάλλον, να μετατρέπει σε πράξη τα ιδανικά τη. Και πρέπει να παραμείνει τέτοιο. Αλλά υπάρχουν μεγάλε ευκαιρίε αν συνδέσουμε τη συνοχή με το κλίμα, με πολύ συγκεκριμένα συγκεκριμένος τρόπος που μπορεί να φέρει αλλαγές στα σπίτια των Ευρωπαίων πολιτών και θα μπορούσαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα στις περιοχές όπου χρειάζεται η πολιτική συνοχή, αλλά και ε, ωφέλει όσον αφορά την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό ήταν ας πούμε ενάμιση σημείο. Δεύτερο τώρα σημείο είναι οι, συνοριακές, οι πολιτικοί μάλλον συνόρων. Ε, δεν ζήτησα συγγνώμη που ε, ε, θίγω ένα θέμα όπου κάναμε πολλά στην περασμένη θητεία. Έχουμε μια μεγάλη δέσμευση με το PDP ώστε να βελτιώσουμε το πώς προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εξωτερικά της σύνορα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει βέβαια να συνοδευτεί και από μια λογική μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη μετανάστευση με το Δουβλίνο ε, και την, ε, το στήριξη του Frontex. Πάντως έχουμε ήδη μαρτυρίες στο διορθωτικό προπολογισμό 4 που αναφέρθηκε νωρίτερα και με τις απαντήσεις που δώσαμε, θα δώσουμε στον επόμενό μας γενικό προπολογισμό. Είναι ένα πιο περίπλοκο, περίπλοκο συγγνώμη, θέμα από ό,τι μπορεί κανείς να πιστεύει και μάλιστα είναι κάτι που αν αποτύχει τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σωστός έλεγχος ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η διεύρυνση του Frontex θα γίνει με σωστό τρόπο, θα αποδώσει αυτό που θέλουμε και δεν θα μετατραπεί σε φιάσκο. Ε, δηλαδή να υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο σχέδιο για το τι κάνει αυτός ο οργανισμός. Μέχρι στιγμής πρέπει να πω ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και τρίτος τομέα που δεν θα σα εντυπωσιάσει ε, είναι το Brexit. Και αν και έχουμε αλλαγή του τοπίου για αυτό το θέμα που ελπίζω πως θα αλλάξει σημαντικά άλλαξαν πολλά πράγματα από το που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Πολλοί πιστεύαμε ότι δεν θα ήμασταν πια εδώ σήμερα, αλλά εδώ είμαστε. Ίσως να χρειαστεί να επανέλθουμε και να επαναξετάσουμε πάλι και, κι άλλο το θέμα αυτό. Ελπίζω πως θα το κάνουμε αλλά ας υποθέσουμε ότι ο σύντομα ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει μια καλύτερη σχέση με αυτό το θέμα από ότι η σχέση που είχε με την αλήθεια μέχρι στιγμής και ότι θα κάνει αυτό για το οποίο λέει και δεν πιστεύω ούτε στιγμή πως θα το κάνει αυτό χωρίς συμφωνία ε, εξόδου. Χρειάζεται λοιπόν συμφωνία εξόδου στο εγγύηση μέλλον, εγώ θα έλεγα πάντως πως δεν πρόκειται προς, προς τα τέλη του 2020 και αν θα γίνει αυτό. Πάντως θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε αν και εφόσον υπάρξει αυτή η συμφωνία και πώς αυτή θα επηρεάσει τον προπολογισμό και η επιρροή αυτή δεν θα φανεί από την πρώτη μέρα αλλά θα φανεί σιγά σιγά ε, με το πέρασμα του χρόνου. Θα πρότεινα λοιπόν να υπάρχει τακτικός και διαρκής έλεγχος εάν γίνει κάτι τέτοιο. Να μην, ε, επίσης να μην σέρνονται αυτές οι επιτροπές με το απότερο μέλλον, αλλά να έχουν ημερομηνία λήξης. Ευχαριστώ. Πεκαρίν. Mr. I'm very new. Είμαι πολύ καινούριος εδώ, Πρόεδρε, στο Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή. Και μάλιστα είμαι ένα πληρωματικό μέλος. Αλλά αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας. Η πρώτη μου ερώτηση είναι άκουσα τα σχόλιά σας και έχω την εντύπωση ότι έχετε κάποιες ανησυχίες ότι ίσως το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεκτεί όλες τις πολύ σημαντικές προτεραιότητες που θέτουμε εμείς ε, εδώ στο Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή. Συμφωνώ με τα όσα είπατε. Το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τα σχολιά μας. Όμως, θα ήθελα να ακούσω εδώ κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές για ζητήματα που σας ανησυχούν ιδιαίτερα. Γιατί σας θέτω αυτό το ζήτημα, γιατί σας το ζητώ. Γιατί ήμουν μέλος ε, του Συμβουλίου πολλά χρόνια και διατέλεσα και υπουργό στην προηγούμενη προεδρία μας. Και θυμάμαι ότι συζητούσαμε τις απόψεις του Κοινοβουλίου και τις λαμβάναμε υπόψη. Και πιστεύω ότι και αυτή τη φορά η φιλανδική κυβέρνηση θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή που ακολουθήσαμε και πριν τόσα πολλά έτη. Αν κάποιος μπορεί να απαντήσει, ευχαριστώ να ακούσω για αυτές τις ε, ιδιαίτερες ανησυχίε ε, που έχουμε. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Κόρμαν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που είμαστε μέλη στην Επιτροπή, λέει ο κύριος Κογμό, και είμαστε ε, πραγματικά αποφασισμένοι και ε, στεναρά απέναντι στο Συμβούλιο για να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο ως Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν για την κλιματική αλλαγή κλπ. Θα ήθελα όμως να αναφέρω κάτι ακόμα, ένα σημαντικό θέμα κατά τη γνώμη μου και για την ομάδα μας του Renew Europe στις διαπραγματεύσεις ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κάνουμε εκτόσεις στις ευρωπαϊκές αξίες. Αγωνιζόμαστε για αυτές, λέει ο κ. Κέρνερ, και θα πρέπει και στο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να φαίνεται. Αυτή είναι θέση της ομάδας μας, αλλά είναι και μεγάλη ευκαιρία στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να προωθήσουμε τα θέματα. Και τελικά, όταν βρεθούν τα χρήματα θα υπάρχουν και, ή μάλλον όταν πρόκειται για τα χρήματα θα γίνουν και μεγάλες μετατοπίσεις ανάλογα με τα θέματα. Και προσβλέπω σε αυτή τη μάχη που πρέπει να δώσουμε ευχαριστώ. Η κυρία Γκέις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με πολλά σημεία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε για το κλίμα, για τους πρόσφυγες, το κράτος δικαίου και φυσικά ε, ένα ισχυρό ρόλο ε, του Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο με αυτοπεποίθηση. Θέλω να αναφέρω ακόμα ένα θέμα που στο παρελθόν δεν ήταν τόσο δημοφιλές αλλά στο μέλλον ελπίζω να έχουμε την υποστήριξή σας και αυτό είναι το gender budgeting, δηλαδή να είμαστε βέβαιοι ότι άνδρες και γυναίκες επωφελούνται εξίσου από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία εμείς ορίζουμε. Είναι ε, χρήματα όλων των φορολογουμένων ανδρών και γυναικών. Και αυτό δεν το επιτάσσει μόνο η δικαιοσύνη, αλλά και η αποτελεσματικότητα των κοινωνιών μας. Να σας δώσω ένα σύντομο παράδειγμα το είδαμε και ε, στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς ότι αυξάνονται τα κονδύλια για την έρευνα, για το Horizon. Αν δίνετε την έρευνα που γίνεται για ασθένειες, ε, τα φάρμακα που απευθύνονται σε γυναίκες δεν διχάνουν σωστής έρευνας. Ε, ας πούμε σε τροχέα σκοτώνονται περισσότερο γυναίκες γιατί οι δοκιμές δεν γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, δεν γίνονται πολλές έρευνες και θα πρέπει να ε, επιληφθούμε. Και χαίρομαι που η κυρία Φόντερ Λάιεν εξήγηλε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι μισή-μισή άνδρες-γυναίκες και αυτό σίγουρα θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει και εμείς να βάλουμε εκεί το λιθαράκι μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ. Κυρία Μάρκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ καταρχήν να πω ότι πρώτη φορά απευθύνομαι στην Επιτροπή, να χαιρετήσω λοιπόν όλους τους παρόντες και τα μέλη της Επιτροπής. Θέλω να θέσω τρία ζητήματα ή να αναφέρω επιχειρήματα για τρία ζητήματα που αναφέρθηκαν εδώ. Καταρχήν, έχουμε το θέμα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Πιστεύω ότι αυτή η προβληματική στη συζήτηση για την ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε μια διάσταση που υπερεύει το θέμα της ε, συμμετοχής ε, στην πρόταση της ε, Κομισιόν για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το κλίμα. Πράγματι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στις προκλητικές εκστρατείες το θέμα του κλίματος έλαβε μια ε, τεράστια θέση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Πορτογαλία μάλιστα. Και η κυρία Φόρτερ Λάιεν στην ε, ομιλία της ε, ανέφερε το θέμα της ένταξης του κλίματος ως συνιστόσα του πολυμετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εγώ θα ήθελα να στραφώ τη συνάδελφο για τις αποκαλούμενες νέες πολιτικές. Γιατί μπήκα στον προπολογισμό σε αυτή την πρόταση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου εις βάρος κυρίως των κονδυλίων συνοχής και επομένως η διάσταση αυτή του κλίματος ε, δεν μπορεί ουσιαστικά να ελοποιείται σε βάρος των κονδύλιων συνοχής. Άλλο θέμα, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Εδώ μιλήσαμε για το θέμα της Frontex και για τη συνεργασία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική ως προτεραιότητα. Όμως εγώ θα ήθελα να ξαναθέσω αυτό το θέμα εδώ ως προτεραιότητα για τα επόμενα πεντέτη. Γιατί εμείς μιλάμε για τη Frontex, για την ένταξη, για μια σειρά ε, διαστάσεων που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό, με το προσφυγικό, με το κλίμα. Και Πράγματι, εμείς θα πρέπει να αξιολογήσουμε διαφορετικά τη διάσταση αυτή, δηλαδή τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Η Πορτογαλία θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου στο πρώτο εξάμεινο του 2021 και θα δέσει αυτό το θέμα ως προτεραιότητα της Προεδρίας και νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει και προτεραιότητα εδώ στη συζήτηση στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Όλμπριχτ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Νομίζω ότι και η κυρία Καρπασάλ έκανε κάποια σχόλια και ήθελα να αντιδράσω πολύ σύντομα γιατί έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας στη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια ευρεία πλειοψηφία συμφωνεί ότι χρειαζόμαστε νέες προτεραιότητες όπως ε, έλεγχος ε, στα σύνορα, κοινό σύστημα σύλλου και άμυνα. Σε αυτά συμφωνούμε. Συμφωνούμε στις μεγάλες προτεραιότητες, ε, στο θέμα του κλίματος, στο να μπει στον προπολογισμό το θέμα του φύλου. Αυτά είναι συμπεφωνημένα από το Κοινοβούλιο. Δεν συμφωνήσαμε όμως με το Συμβούλιο στα εξή. Καταρχήν, για το ποσό στον προϋπολογισμό. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφωνία εκεί, αλλά είναι μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αλλά ακόμη περισσότερο μεταξύ των κρατών μελών εντός του Συμβουλίου. Το γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία εντός του Συμβουλίου. Γι' αυτό προσπαθήσαμε για πρώτη φορά να κάνουμε την εξή ανάλυση. Πόσο θα κοστίσουν οι προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί από τα κράτη-μέλη και κάνουμε την ανάλυση αυτή και το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι 1,3 ε, του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος. Ε, ενώ ε, η ανάλυση συμβουλίου ήταν 1% τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν ήταν 1,08 χωρίς το ειδικό ταμείο. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου που έχει ψηφιστεί από την ευρία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Δεν συμφωνήσαμε ότι οι νέες προτεραιότητες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τις παλιέ πολιτικές. Δηλαδή να αφαιρέσουμε χρήματα από τη γεωργία και τη συνοχή και να μεταφέρουμε κονδύλια στις νέες προτεραιότητες. Σε αυτό δεν συμφωνήσαμε. Είπαμε εντάξει, θέλετε νέες προτεραιότητες, εντάξει, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Το άλλο θέμα είναι το θέμα τη ευελιξία. Αν θα πρέπει να είναι ευέλικτο ο προπολογισμό ή όχι. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να μειώσουν αυτή την ευελιξία στο μηδέν. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ο ρόλο του Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Δηλαδή, διάμεση αναθεώρηση ε, ή ανασκόπηση. Ε, και υπάρχει διαφωνία και σε αυτό, γιατί δεν θέλουν κάποια κράτη-μέλη να υπάρχει καθόλου τέτοια ενδιάμεση ε, ανασκόπηση, μόνο ενδιάμεση αναθεώρηση. Έτσι λοιπόν, συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο για τις νέες προτεραιότητες, αλλά διαφωνήσαμε σε ό,τι αφορά τη δομή και τα ποσά. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, τώρα τι έχουμε επιτάπητος. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε τις προτάσεις της Κομισιόν από το Μάιο του 2018 Έχουμε πολλές προτάσεις του Κοινοβουλίου. Η τελευταία είναι από την ενδιάμεση έκθεση του Νοεμβρίου 2018 και αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε από μια μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Και παρατηρούμε τι συμβαίνει τώρα στο Συμβούλιο. Γιατί η Φιλανδική Προεδρία προσπαθεί τώρα να καταλήξει με κοινή θέση με τα κράτη-μέλη. Αυτά τα έγγραφα, λοιπόν, ε, έχουμε τα έγγραφα Κομισιόν Κοινοβουλίου και περιμένουμε του Συμβουλίου. Και να είμαι κάπως προκλητικός, μια πρόταση βάσει της δικής μου εμπειρίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον τι θα γίνει με τη νέα Κομισιόν. Γιατί θα αναλάβει καθήκοντα η νέα Κομισιόν, θα έχουμε τις ακροάσεις. Δεν είναι μια ερώτηση στην Κομισιόν, μια δήλωση είναι απλώς. Πραγματικά με ενδιαφέρει να δω αν η νέα Κομισιόν θα τηρήσει όλα όσα υπάρχουν στα έγγραφα της Κομισιόν του Μαΐου 2018. Γιατί αυτά είναι απολύτως βασικά. Φυσικά, αν διατηρήσουμε την ίδια θέση με τον Νοέμβριο του 2018, θα το δει αυτό και το Συμβούλιο. Όμως, έχουμε το Ταμείο Γιούνκερ, το σχάλι, που εμφανίστηκε μετά την απόφαση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και άλλαξε εντελώ όλη τη δομή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ρωτήσουμε τους νέους επιτρόπους υποψηφίου, Τι θα γίνει με το πολιτές στην Θέλετε να το διτηρήσετε ω έχει, θέλετε να το αλλάξετε. Γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το κοινοβούλιο. Είναι κάπως προκλητική αυτή η ερώτηση πριν από την εκλογή των νέων επιτρόπων, αλλά δεν θα πρέπει να την ξεχάσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Όλμπριχτ. Άλλα σχολεία υπάρχουν. Ή θέλετε να πείτε κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ζωντανή συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Να υπενθυμίσω ότι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός δεν είναι απλά ένα σύνολο δεδομένων και αρνητικών στοιχείων, αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες και διαμορφώνει την κατεύθυνση προ την οποία οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν προφανώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεργά θα πρέπει να συμμετέχει και προδραστικά. Ένα προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί καλά θα πρέπει να παράγει αποτελέσματα και πάνω απ' όλα προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, τους φορολογουμένου. Επομένως, ενώ θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τις κύριες εργασίες μας, θα ήθελα να βρούμε χρόνο στις ημερήσεις διατάξεις της Επιτροπής μας για να έχουμε και γενικές συζητήσεις για νέα ζητήματα που εμφανίζονται και που έχουν αντίκτυπο δημοσιονομικό ή άμεσο ή ενδυνάμει. πρώην Υπουργό Οικονομικών σας διαβεβαιώ ότι αν δείτε προσεκτικά κάθε ε, θέμα τελικά έχει δημοσιονομικό αντίκτυπο άμεσα ή έμεσα. Και φυσικά ανυπομονώ να συζητήσω περαιτέρω μαζί σας ε, αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ. We can go to... Προχωρούμε λοιπόν τώρα στο σημείο 10. Κτηριακή πολιτική. Αύριο θα το συζητήσουμε για την ψηφοφορία, μάλλον γιατί πρόκειται για κάτι που χρειάζεται πρώτερη έγκριση. Κανονικά θα πρέπει να περάσουμε στο σημείο 11, όπως γνωρίζετε μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών και έχει προβλεφθεί να αρχίσει ακριβώς σε μία ώρα από τώρα, στις 5.30. Προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, να διακόψουμε και να τα ξαναπούμε στις 5,5 όπως είχε προβλεφθεί. Για το Ταμείο Μαντάτ. Αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ. AUTHORWAVE Ε. Καλησπέρα σας και πάλι. Προτείνω να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας με το σημείο 11. Καλωσορίζω τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών, ιδιαίτερα τον πρόεδρο κύριο Βαζικόφσκι. Το θέμα αφορά την επέκταση του καταπιστευματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για απάντηση στη Συριακή κρίση. Το Ταμείο Ματάντ είναι η δεύτερη φορά ε, που σε συνεργασία με άλλη επιτροπή, η επιτροπή μας καλείται να ε, γνωμοδοτήσει για την επέκταση του Ταμείου και παράταση μέχρι το ε, Δεκέμβριο του 2020. Στο παρελθόν είχαμε εκφράσει έντονες επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα διάφορα καταπιστεύματα ε, ρήμην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χρησιμοποιούνται αυτά τα ταμεία παράλληλα με τα κρατημέλη και άλλους δωρητές. Στο άρθρο 234 ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός εκφράζει αυτή τη δυσφορία και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο σχέδιο ε, πρότασης για ίδρυση τέτοιων ταμείων ή για παράταση τους για δράσεις ε, κατεπήγουσης ή μετά από ε, ε, Να ζητάει τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα συνεδριάζουμε μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών και θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Βασικόφσκι. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή είναι δύσκολο το όνομά μου, πολωνικό. Θα έχετε πέντε χρόνια για να το μάθετε. Μην ανησυχείτε, θα τα λέτε τέλεια σε πέντε χρόνια. Θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του Προέδρου μας, David McAllister, της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Είναι με μια ειδική αποστολή για να παρατηρήσει τις εκλογές στην Ουκρανία. Εργάζεται πολύ σκληρά. Είχα την ευκαιρία να διαβάσω τις εκθέσεις του ε, και τις δηλώσεις του και πιστεύω ότι θα μάθουμε περισσότερα για την κατάσταση στην Ουκρανία και τα αποτελέσματα των εκλογών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών την Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ που έχω την ευκαιρία για πρώτη φορά να συμπροεδρεύω σε αυτή τη σημαντική κοινή συνεδρία των Διεπιτροπών μας. Όπως είπε ο συνάδελφο, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια πρόταση με αιτιολόγηση για ποιο λόγο θέλει επέκταση, παράταση του ταμείου αυτού. Δεν θέλω να προεξοφλήσω εγώ τις, ή να αποτρέξω ε, τις εξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί την κατάσταση στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή με μεγάλη ανησυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να υποστηρίξει τις χώρες που πλήττονται από την Συριακή κρίση, ιδιαίτερα τις γειτονικές χώρες. 5,6 εκατομμύρια πρόσφυγες, ίσως και περισσότεροι, ε, ε, ζουν σε γειτονικέ χώρες. 5,6 εκατομμύρια είναι καταγεγραμμένοι σε χώρες όπως είναι ο Λίβανος, η Ορδανία, η Τουρκία και το Ιράκ. Και εδώ στην Ευρώπη φυσικά έχουμε ε, πρόσφυγες και μετανάστες. Το Ταμείο Μαντάτ είναι το βασικό ταμείο που υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τις χώρες που τις υποδέχονται μαζί με τη βοήθεια για την Τουρκία. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση κατέληξε η αξιολόγηση ότι είναι πολύ αποτελεσματική η λειτουργία του καταπιστεύματος αυτού και έχει παράξει και προστιθέμενη αξία. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί και κάποιες αδυναμίες και έχουν γίνει συγκεκριμένες συστάσεις. Θα μας ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να δώσει συνέχεια σε αυτές τις συστάσεις και τις επισημάνσεις. Επίσης θα θέλαμε ή δυνατό να μας επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Ταμείο δεν θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση της Συρίας, εκτός αν υπάρχει σαφής δέσμευση από το καθεστώς Ασάντ ότι σέβεται τη διαδικασία της Γενέβης και καταλήξει σε μια πολιτική λύση που θα τερματίσει τη σύρεξη και θα υπάρξει μετάβαση ε, στη Συρία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ποπόφσκι, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΑ, να μας παρουσιάσει ε, το αίτημα επέκτασης και παράτασης της λειτουργίας του ε, καταπιστεύματος Μαντάντ. Επίσης, να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη Συρία κατά αυτόν τον τρόπο μετά το 2020. Θα κάνω και την πρώτη ερώτηση λοιπόν ο Συμπροέδρος πριν την παρουσίαση. Κύριε Ποπόσκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο προέδρους. Ευτυχώς είναι κάπως πιο εύκολο να προφέρει κανείς το όνομά μου, αλλά και πάλι πολωνικό. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, όπως είπε και ο κύριος Βασικόφσκι να περιγράψω την κατάσταση. Υπάρχει συνεχής ανάγκη για την δική μας υποστήριξη. Η κρίση στη Συρία δεν έχει τελειώσει και ούτε πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Εκατομμύρια άνθρωποι και πρόσφυγες αλλά και κοινότητες φιλοξενίας στις γειτονικές χώρες χρειάζονται την υποστήριξή μας γιατί η κρίση και η διάρκειά της έχει μεγάλο αντίκτυπο στις εθνικές αρχές. Επίσης, θα απαντήσω αμέσως στην πρώτη ερώτηση, όσο δεν υπάρχει πολιτική μετάβαση στη Συρία, δεν πρόκειται να δεσμευτούμε στην ανοικοδόμηση. Θα συνεχίσουμε με κάποια πολύ συγκεκριμένη ανθρωπιστική στήριξη εντός της Συρίας, αλλά δεν θα υπάρξει ανοικοδόμηση εκτός αν υπάρξει πολιτική μετάβαση και εκτός αν οι συνθήκες ε, για να υπάρχουν εκούσιες επιστροφές που να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όμως ε, δυστυχώς αυξάνεται η πίεση στις ε, χώρες φιλοξενίες. Υπάρχει μια ρητορική κατά των προσφύγων, κυρίως στο Λίβανο, με περίπτωση που έχουμε, περιπτώσεις έχουμε καταστροφή ε, κάποιων καταφυγίων προσφύγων ε, και ιδίω βλέπουμε στο Λίβανο να συμβαίνει αυτό, λίγο λιγότερο στην Ιορδανία και στην Τουρκία, αλλά δυστυχώ υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Το καταπίστευμα Μαντάντ έχει υποστηρίξει πάρα πολύ του πρόσφυγε και τι κοινότητε υποδοχή και έχει αποφύγει στο να αποφευθεί μια κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάρρευση στην Ιορδανία και τον Λιβανό. Έχουμε φτάσει στο 1,8 δισεκατομμύρια με το 1,6 δισεκατομμύρια του προπολογισμού να έχουν ήδη καταναμηθεί σε δράσεις και το 1,3 να έχουν τύχει ε, σύμβαση σε διάφορα project. Ε, φτάνουμε σχεδόν στο στόχο των 1,7 που τέθηκε το 2015. Προέρχονται τα κονδύλια, κυρίως από το κράτη-μέλη είναι το 18% και ένα 10% του προπολογισμού όσο έχει σήμερα. Έχουμε συστήσει ένα σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης. Οι αποδείξεις μας δείχνουν ότι το καταπίστευμα είναι αποτελεσματικό εργαλείο που μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά μεγάλα προγράμματα και μας παρουσιάζει αποτελέσματα καλής ποιότητας. Τα αποτελέσματα που συλλέχθησαν στις τριμηνίες εκθέσεις μας είναι διαθέσιμα και στην αίθουσα αλλά και επιγραμμικά. Αναφερθήκαμε στην στατική ενδιάμεση εξολόγηση που ζητήσαμε το 2018. Ε, το ε, Ταμείο, το UTF, ε, ήταν αποτελεσματικό εργαλείο και έφτασε σε πολλούς δικαιούχους συγκριτικά με χαμηλό κόστος. Επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει αποτελεσματικά και προσαρμόστηκε στη δυναμική στην περιοχή. Το Καταπιστημονικό Ταμείο δημιούργησε προσθέμενη αξία σε σχέση με μονομένες προσπάθειες από τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν αυτό ε, στις συστάσεις βλέπουμε να παραταθεί το Ταμείο πέρα από το Δεκέμβριο του 2019 προκειμένου να μπορεί ε, να καλύπτει τις ανάγκες των δικαιούχων στις χώρες αυτές. Υπάρχει και συνένεση μεταξύ ε, των μελών του Δικαιωτικού Συμβουλίου ότι συνεχίζει να έχει αξία το καταπιστευματικό ταμείο και ότι θα έπρεπε να ε, μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε στις ανάγκες εκατομμυρίων ανθρώπων στην περιοχή. Στη συνεδρίασή του το Δεκέμβριο, το επιχειρησιακό ταμείο του Trust Fund ομόφωνα ζήτησε από την Κομισιόν να επεκτείνει τη θητεία, να παρατείνει τη θητεία για ένα χρόνο. Συνοδεύτηκε από νέα χρηματοοικονομική υποστήριξη από πολλά κράτη-μέλη. Άλλοι ε, είπαν ότι θα προσφέρουν περαιτέρω στήριξη το 2019 συνεχίζουν να έρχονται εισφορές και από τα κράτη-μέλη και από την τελευταία ε, συνεδρίαση όπου είχαμε δεσμεύσει της ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2019. Ε, τα έχουμε συγκεκριμένα κονδύλια που έχει λάβει το Ταμείο και αν δεν υπάρχει παράταση δεν θα μπορούν να υπογραφούν περαιτέρω συμβάσεις πέρα από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 ούτε να δεσμεύσει τη διαθέσιμα κονδύλια. Έτσι λοιπόν έχουμε πρόκληση σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, διοίκησης. Ε, η Διευθύντρια πιστεύει ότι θα έπρεπε να αρνηθεί επιπρόσθετα κονδύλια για τα οποία έχουν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη και δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί περαιτέρω χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό αν δεν υπάρχει αυτή η παράταση. Έτσι λοιπόν, ε, κατά ένα επιπλέον έτος το UTF θα επικεντρωνόταν στην Ιορδανία και στο Λίβανο και ω ένα βαθμό στο Ιράκ, έτσι όπως συστήνεται στην ενδιάμεση αξιολόγηση, καθώς η Τουρκία καλύπτεται από ένα ξεχωριστό μέσο, από ένα ξεχωριστό μηχανισμό, το μηχανισμό για τους πρόσφυγες για την Τουρκία στο δεύτερο στάδιο θα επικεντρωθούμε στην ενδυνάμωση της αυτάρκειας ε, των προσφύγων και της υποστήριξης των συστημάτων ε, στις ε, χώρες υποδοχής προκειμένου να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, παιδεία, υγεία, διαχείριση αποβλήτων όμως διαφέρει η κατάσταση στις δύο χώρες, γιατί στο Λιβένο είναι σε μικρότερα καταφύγια ζουν πρόσφυγες, όχι σε καταβλισμούς, ενώ στην Ιορδανία πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν σε καταβλισμούς και χρειάζεται λοιπόν μια προσέγγιση πολύ συγκεκριμένη. Τώρα, για την πρώτη σας ερώτηση, Πρόεδρε, για το θέμα της παράτασης. Αυτό εξαρτάται από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είμαστε σε θέση να δεσμευτούμε τώρα, πέρα από το 2021, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί αυτό θα αποτελεί πηγή πρόσθετης χρηματοδότησης, γιατί ακολουθήσει μετά το 2021. Και βεβαίως, στην πρότασή της, η Κομισιόν Εντό του πακέτου του πολιτισμού συνομικού πλασίου, η Κομισιόν προτείνει μια, ένα νέο ε, παγκόσμιο εργαλείο πολιτικής που θα έχει και ένα αποθεματικό κονδυλίων για σχέδια που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αναπτυχθεί αυτό μέχρι τα τέλη του έτου έτσι όπω ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σχόλια παρακαλώ τοποθετήσεις για αυτά που ακούσαμε. Α, συγγνώμη, προηγουμένως θα πρέπει να δώσω το λόγο και στην κυρία Κόμς. Όχι. Όχι. Απουσιάζει. Όχι. Άρα ποιος θέλει να σχολιάσει αυτά που ακούσαμε. Κύριε Γόρδια ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις εξηγήσει. Έχω μια ερώτηση. Εδώ είμαι. Ε, στα δεξιά σας. Εδώ. Παρόλο που μας ενημερώσατε, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ε, για τα καταπιστεύματα έτσι κι αλλιώς, δεν θα σας εκπλήξει. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού ποτέ εμείς δεν αφισβητήσαμε το σκοπό για τον οποίο δημιουργούνται τα ταμεία αυτά, αλλά τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε την εκτέλεση. Το είπε ε, στο παρελθόν και ο πρόεδρος Σαρτοή, ότι ήταν ένας γαλαξίας εκτός του προϋπολογισμού και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να δούμε ε, ποια χρήματα εκταμιεύτηκαν, από πού, πώς συνελέγησαν, για ποια προγράμματα ε, κτλ και πού κατευθύνονται. Αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ το δημοσιονομικό μας έργο. Φυσικά και προφανώς κατανοούμε τους σκοπούς και τον αντίκτυπο που έχει χρήση αυτών των κατεπιστευματικών ταμείων ε, επιτόπου στο Λίβανο, την Ιορδανία και το Ιράκ. Είναι πολύ θετικά. Αλλά από τη σκοπιά του προπολογισμού και της Επιτροπής Προπολογισμών πάντα έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για το πώς μπορούμε να ελέγξουμε την εκταμείευση και την εκτέλεση αυτών των κονδυλίων. Τούτων λεχθένων προτείνεται παράταση μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου. Γιατί, περίεργο, και γιατί όχι στις 31, όπως οποιαδήποτε άσκηση οικονομικό έτος. Και ε, το παρατείνεται μέχρι το 2020 γιατί την 1η Πρώτου του 2021 αρχίζει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί εκτός αυτού. Σε αυτό το νέο Ταμείο Συνεργασίας, πώς θα λέγεται, θα ενταχθεί και ε, το σύνολο των καταπιστευματικών ταμείων και στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχουμε αυτά τα εργαλεία. Έχω και άλλη ερώτηση. Βεβαίως πήραμε ε, έγγραφα, αλλά ήταν λίγο ταραγμένη η αρχή της θητείας. Η παράταση τι σημαίνει. Ο ευρωπαϊκός προπολογισμό θα πρέπει να δώσει περισσότερα κονδύλια. Αν ναι, πόσα και ε, αν το έχετε συμπεριλάβει στην πρόταση ε, του προπολογισμού που κατέθεσε τον Ιούνιο ο κύριος Oettinger για το 2020, γιατί εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα μας κοστίσει χρήματα από τον προπολογισμό αυτή η παράταση ή όχι. Και αν μας κοστίσει, έχει ήδη προβλεφθεί στον προπολογισμό του 2020 και κάτι άλλο σε σχέση με την Τουρκία. Διότι είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει άλλο trust fund. Αν δεν απατώμε όμως, υπάρχουν κάποια έργα που χρηματοδοτούνται από το Μαντάτ και τρέχουν και στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο περίπλοκο είναι να παρακολουθούμε όλες αυτές τις δράσεις, πώς διαφοροποιούνται, πώς συμπληρώνονται και τι διαφορά έχει αυτό που κάνουμε στην Τουρκία από το συγκεκριμένο ταμείο για την Τουρκία και αυτά που κάνουμε από το ταμείο Μαντάτ. Αυτά ε, από ερωτήματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριανή, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καθώς είμαι νέο μέλος και δεν είμαι μέλος ε, της Επιτροπής του Προϋπολογισμού, ε, σας δω και των προτέρων, συγγνώμη αν είμαι λίγο εκτός θέματος. έχω επισκεφθεί τη Συρία έξι φορές τα τελευταία χρόνια και θα ξαναπάω σε τέσσερις εβδομάδες. Ε, τη γνωρίζω λοιπόν αρκετά καλά. Κατάλαβα τη βασική θέση που λέει ότι δεν θα συμμετέχουμε στην ανοικοδόμηση της Συρίας από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει πολιτική μετάβαση. Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή, δεν την αμφισβητώ. Όμως ρωτώ με, αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες πρέπει να περιοριστούμε στους εξωτερικούς πρόσφυγες και συστηματικά να ξεχνάμε τους εσωτερικά εκτοπισμένους. Έχετε δίκιο ότι είναι όλοι αυτοί οι πρόσφυγες στο Λίβανο, στην Ιορδανία και στο Ιράκ, αλλά 5 με 7 εκατομμύρια είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, έχουν είτε φύγει από τις ζώνες που ελέγχει η Τζαμπάτα και είτε από τις ζώνες που ελέγχε ο Νταές. Ε, το θέμα είναι λοιπόν, θέλουμε να είμαστε αποδιωτικοί χωρίς να μπούμε στην ανοικοδόμηση. Δεν μπαίνω, σας είπα, επισέρχομαι σε αυτό το θέμα, αν και δεν είμαι της ίδιας άποψης. Θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς, γιατί έχουμε οργανώσεις όπως ε, η Ερυθρέα ε, Έλληνος ή άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν αποτελεσματικά στη Συρία χωρίς αναγκαστικά να περνάμε από την κυβέρνηση. Στο περασμένο Νοέμβριο επισκέφθηκα την Ντούμα στην Ανατολική Γκούτα. 500.000 πρόσφυγες που ζουν σε δραματικές ε, ε, συνθήκες. Στο Αλέπ έφτασα μία εβδομάδα μετά την πάυση των εχθροπραξιών. Και εκεί ε, δράμα η Ευρώπη, αν θέλουμε να έχει θετική εικόνα, κάτι πρέπει να κάνουμε πέρα από τις πολιτικές επιλογές. Πιστεύω πως μπορούμε να δράσουμε προς τους πρόσφυγες που παραμένουν εντός της Συρίας. Καταρχάς γιατί είναι καλύτερα να μείνουν στη Συρία παρά να πάνε στους γείτονες ή να έρθουν στην Ευρώπη και γιατί είναι επίσης το καλύτερο στάδιο για να μπορούμε να διευκολύνουμε μια επανεγκατάσταση. Και να θυμίσω κάτι ακόμα. Η Συρία σήμερα ε, είναι υποκυρώσεις όσον αφορά το ιατρικό υλικό και τα φάρμακα. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε κάπως καλύτερη μεταχείριση των προσφύγων, όταν μπαίνει κανείς στη Συρία βλέπει, και έχω και φωτογραφίες για όσους ενδιαφέρεστε, βλέπουμε ε, ε λίστες από υλικό, σκάνερ, υλικό εργαστηρίου που δεν λειτουργεί πλέον γιατί απλούστατα μπλοκάρεται η παράδοση εξαρτημάτων, ανταλλακτικών για επισκευές. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε εκεί να ενεργήσουμε. Καταλαβαίνω τα εμπάργο για το υλικό κτλ. Αλλά το να μπλοκάρει κανείς την επισκευή ενό σκάνερ δεν πιστεύετε ότι στην πραγματικότητα στην ουσία τιμωρεί όλο τον πληθυσμό. Ε, το ερώτημά μου είναι απλό λοιπόν. Αυτό το, το, ταμείο μπορεί να επεκταθεί και στους εσωτερικά εκτοπισμένους Σύριους που είναι και οι πιο πολλοί άριθμοι. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια. <clears throat> Ε, καλημέρα σας. Ε, ονομάζομαι Φαμπιέν Κέλλερ και δεν έχω πια φωνή. Λυπούμαι γι' αυτό. Ε, ε, είμαι νεοεκλεγμένη από την ομάδα Renew από τη Γαλλία και έχω κάποιες βασικές ερωτήσεις. Μήπως ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μπορεί να μας δώσει κάποιες τάξει μεγέθου, για, μεγέθους για τις άλλες χρηματοδοτήσει, ας πούμε για τα Ηνωμένα Έθνη, άλλα αναπτυξιακά ταμεία, για να έχουμε μια ιδέα του ποιο κομμάτι καλύπτει αυτό το ταμείο Μαντάτ, το καταπίστευμα σε σχέση με τη διεθνή προσπάθεια. Και επίσης, μπορείτε να μας δώσετε ποιο είναι το νούμερο για την Τουρκία για να μπορούμε επίσης να συγκρίνουμε, αφού κατάλαβα ότι πρόκειται για ξεχωριστό καταπίστευμα. Τώρα όσον αφορά τις αρμοδιότητες ίσως της ΑΦΕΤ. Τι γίνεται με τη ζωή στα καταβλισμούς, την επιβίωση των προσφύγων και σε αντίθεση με την, τα όσα θα δοθούν για νοικοδόμηση ή για επιστροφή. Κοιτάξτε, ο κλιματισμός του Ευρωκοινοβουλίο θα με αποτελειώσει, δεν... Ναι. Υπάρχουν επίσης ιδέες γιατί εδώ ανανεώνουμε για ένα χρόνο. Έχουμε μια ιδέα για το ποιες είναι οι προοπτικές για αυτό το ταμείο που θα περιληφθεί στις ε, πολυετής προπτικές. Πάλι είναι περισσότερο θέμα της ΑΦΕΤ όσον αφορά τις ανάγκες και τον τρόπο παρέμβασης και τις δημοσιονομικές ανάγκες που συνδέονται με, με αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Όλμπριχτ, μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως μέλος της Επιτροπής Προπολογισμού έχω μια ερώτηση σε σχέση με τον προπολογισμό και τις προπτικές, διότι Ανέκαθεν στην Επιτροπή Προπολογισμού υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με αυτά τα καταπιστεύματα και σε ποιο βαθμό αυτά ελέγχονται από το Κοινοβούλιο ή όχι, αν είναι ανεξάρτητα, αν είναι εκτός του προπολογισμού, εντό του προπολογισμού κτλ. Αλλά εάν θέλουμε να παρατείνουμε την κατάσταση. Τι είναι, ποια είναι η αναμενόμενη δομή του καταπιστεύματος για το μέλλον. Τι γίνεται με τις αποφάσεις των συγκεκριμένων κρατών μελών να συμμετέχουν τους επόμενους μήνες και χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ποιο ποσοστό είναι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό και ποιο ποσοστό είναι των κρατών μελών. Γιατί όταν, αρχίσαμε, όταν αρχίσουμε να συζητάμε το PDP θα είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό γιατί ε, Ποια είναι τα ποσοστά λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι κρατών μελών είναι σταθερό ή κάθε χρόνο εξαρτάται από τις πολιτικές αποφάσεις των κρατών μελών. Ποια είναι η δομή αυτού του ταμείου καταπιστεύματος. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Κύριε Σεράνκα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του ECR εγώ υποστηρίζω τα όσα είπαμε μέχρι τώρα. Η δική μου παρέμβαση προκύπτει από την έκθεση που λέει ότι το δράμα στη Συρία κάπως βλύνεται με αυτές τις παρεμβάσεις. Είναι θετική η συμβολή της Ένωσης. Όμω έχω να κάνω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Από ό,τι κατάλαβα από αυτέ τις πρώτες επαφέ για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το καταπίστευμα αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στην πολιτική για τη μετανάστευση. Αυτή είναι η κατεύθυνση από ό,τι κατάλαβα της Κομισιόν. Άλλες ερωτήσεις. Μάλιστα, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια άλλη ερώτηση όσον αφορά τους ε, πρόσφυγες εντός Συρίας. η μελλοντική, το μελλοντικό καθεστώς για την Βόρεια Συρία φαίνεται να είναι ακαθόριστο αυτή τη στιγμή. Ε, μπορείτε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Έχω και εγώ να ρωτήσω κάτι. Διότι το Κοινοβούλιο εκτιμά πολύ το γεγονός ότι καλείται στις συνελεύσεις ε, του Διοικητικού Συμβουλίου, όμως στο παρελθόν οι ημερομηνίε δεν ε, ε, μας φόλεψαν. Δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε. Μήπως μπορείτε να λάβετε υπόψη το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου όταν ορίζετε τις συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Καταπιστεύματος. Αυτά και θα δώσω το λόγο βέβαια στον εκπρόσωπο της Κομισιόν γιατί ετέθησαν πολλά συγκεκριμένα ερωτήματα. Thank you very much. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Καταρχήν, να απαντήσω με τη σειρά οι ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Το συζητάμε αυτό εδώ και καιρό. Σωστά αναφερθήκατε στην ανταλλαγή με τον Επίτροπο Έτιγκερ και έρχομαι κατευθείαν στην ερώτηση του Πρόεδρου. Ήταν ένα πρώτο βήμα, αλλά χρήσιμο να κληθούν οι ευρωβουλευτές σε όλα τα συμβούλια όλων των καταπιστευμάτων και της Διευθύνουσας Επιτροπής του Μηχανισμού για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία Παραδέχομαι ότι κάναμε κάποια στιγμή λάθο, γιατί βάλαμε τη συνεδρίαση κατά εβδομάδα Στρασβούργου. Αλλά δεν θα ξαναγίνει. Θα διασφαλίζω πάντα ότι θα γίνεται εβδομάδα όταν θα είναι οι ευρωβουλευτέ τη Βρυξέλλε. Και βεβαίω ε, με χαρά ε, θα δω τα μέλη που έχουν επανακλογεί στι αντίστοιχε επιτροπέ να παραβρεθούν στις συνεδριάσεις. Επίσης, στο παρελθόν, μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, αλλά και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, πήγαν ε, σε σε αποστολές επιτόπου για να δουν τα διάφορα προγράμματα και σχέδια επιτόπου και ευχαρίστως θα διευκολύνουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Βεβαίως, το Trust Fund ε, σήμερα είναι εκτός προϋπολογισμού και αυτό σχετίζεται με τις διατάξεις του, του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Όπως σας είπα, ε, αυτό στο μέλλον εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθούν και τι μορφή θα πάρουν διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς προτείνουμε να έχουμε ένα εργαλείο που να καλύπτει τα πάντα, τη γειτονία, την ε, διεθνή συνεργασία δηλαδή τη διαχείριση στο μεταναστευτικό και την απάντηση στην κρίση και κατόπιν η Δημοσιονομική Αρχή θα ήταν αρμόδια να αποφασίσει κάποια στιγμή αν ε, τα τραστφάν, τα θα συνεχίσουν να τρέχουν παράλληλα ή όχι. Εμείς είχαμε τη λογική να προτείνουμε ένα εργαλείο εντός του προπολογισμού που θα κάλυπτε όλες τις ανάγκες που καλύπτονται από τα καταπιστεύματα τώρα. Βέβαια, ερχόμαστε στο θέμα της οικονομική βιωσιμότητα και πόση χρηματοδότηση θα ήταν διαθέσιμη, αλλά θα επανέλθω στη συμμετοχή των κρατών μελών σε λίγο. Εντός της Συρίας. Όχι. Για τον προπολογισμό για το 2020 δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποια τελική μορφή θα πάρει η δημοσιονομική διαδικασία. Προτείνουμε μία συνεισφορά 150 εκατομμυρίων αυτό συνάδει με την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μάρτιο του 2019. Η σχέση μεταξύ του Μαντάντα και του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία είναι κάπως πολύπλοκη, γιατί το Trust Fund προηγείται του μηχανισμού, έτσι λοιπόν το καταπίτασμα πρώτα συστάθηκε, κατόπιν είχαμε το μηχανισμό μετά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του Μαρτίου 2016. Επομένως, ε, μία σειρά δράσεων στην Τουρκία που στοχεύουν στον ε, πληθυσμό της Συρίας ξεκίνησαν υπό το Trust Fund και μπορούμε να αποβλακούμε στο μέλλον γιατί έχουμε ένα ξεχαριστό μηχανισμό γι' αυτό δράσεις εντός της Τουρκίας υπό το καταπίστευμα φτάνουν ακόμη στο 31% για να είμαι Έτσι λοιπόν ο συνολικός προϋπολογισμός είναι τώρα 1 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια και λιγότερο από το 1 τρίτο δεσμεύεται στην Τουρκία. Ουσιαστικά έχουμε μια διασταυρούμενη δράση μεταξύ του Μαντάντ και του Μηχανισμού για την Τουρκία. Τέθηκε και μια άλλη ερώτηση. Ο συνδυασμένο προπολογισμό για το μηχανισμό είναι 6 δισεκατομμύρια. Το συμφωνήθηκε το Μάρτιο του 2016. 3 δισεκατομμύρια στην πρώτη δόση και στη δεύτερη δόση πάλι 3 δισεκατομμύρια. Την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν υιοθέτησε μια τελική οικονομική απόφαση με την οποία δέσμευσε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη δόση. Δηλαδή η χρηματοδότηση τώρα έχει διασφαλιστεί για τη δεύτερη δόση, αλλά φυσικά αυτό πάλι τρέχει μέχρι το 2021 και πάλι. Δεν συζητάμε κάποια παράταση στο μέλλον του μηχανισμού για την Τουρκία γιατί συνδέεται και με τις ε, δυνατότητες χρηματοδότησης ε, εντός του μελλοντικού πολίτες δημοσιονομικού πλαισίου και είναι ακόμη πολύ νωρί. Για τις δραστηριότητες εντός της Συρίας και συγκεκριμένα τις δραστηριότητες που προσθέτουν τους εσωτερικά εκτοπισμένους. Όπως είπα, στη Συρία αναλαμβάνουμε δράση μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων όπως ο αλλά φυσικά έχουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ τη ε, δουλειά παραδοσιακή ανάπτυξη όπω ε, τη ανοικοδόμηση που δεν γίνεται και τη ανθρωπιστική ε, δουλειά που συνεχίζεται. Έτσι λοιπόν οι συνάδελφοι από την ΕΚΟ είναι ενεργοί εκεί και ο προπολογισμό είναι 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Αντιμετωπίζουν λοιπόν πάρα πολλέ δυσκολίε πρόσβαση στου δικαιούχου πρέπει να συνεργάζονται με κυβερνητικούς οργανισμούς, πάντοτε είναι δύσκολο αυτό. Και κάποιοι τέτοιοι οργανισμοί ε, είναι στον κατάλογο κυρώσεων του ΟΗΕ, έτσι λοιπόν αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. σε τη σχέση, το επίπεδο χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμο για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, 3 συν 3 δις ευρώ σε ό,τι αφορά τώρα τους άλλους δωρητές, τον ΟΗΕ, οι διμερείς δωρητές, δεν έχω τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά μπορώ να σας δώσω γραπτές πληροφορίες. Για τα Ηνωμένα Έθνη μπορεί να είναι κάπω πολύπλοκο γιατί εμεί στη Συρία χρηματοδοτούμε πολλέ από τι δράσει του ΟΗΕ. Στη Συρία, ένα από του κύριου εταίρου μα στην Τουρκία είναι με χάρη το πρόγραμμα του ΟΗΕ για το περιβάλλον. Με χάρη έχουμε και τη UNICEF με την οποία συνεργαζόμαστε και πολλού άλλου. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη δομή του Ταμείου Καταπιστεύματος και το επίπεδο των εισφορών των κρατών μελών. Καταρχήν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ όλων των Trust Fund και του μηχανισμού για τις πρόσφυγες στην Τουρκία. Ο μηχανισμός είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και της τουρκικής κυβέρνησης. Και δυνάμει της συμφωνίας, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να συνεισφέρουν στο μηχανισμό έτσι λοιπόν εγώ ως πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής ε, είμαι ο παραλήπτης αυτών των πιστοποιητικών εισφορών. Είναι υποχρέωση λοιπόν. Ενώ όλες οι εισφορές για τα καταπιστεύματα είναι ακούσεις. και εδώ ξεκινά το πρόβλημα προς στιγμή. Οι εισφορές των κρατών είναι περίπου το 10% του προϋπολογισμού του Μαντάντ. Δεν είμαι σίγουρος τι γίνεται σε άλλα καταπιστευματικά ταμεία, αλλά μάλλον είναι παρόμοιε συνολογίε. Συνεχίζουμε να απευθύνουμε έκκληση για πρόσθεσει φορέ, για τη Συρία, για το καταπίστευμα για την ε, Βορεια αλλά φυσικά είμαστε στα χέρια των κρατών μελών, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη χρηματοδότηση και την πολιτική του βούληση. Επομένω, δεν μπορώ να προβλέψω αν είναι σταθερή αυτή η και μπορεί να ακολουθεί στο μέλλον. Μόνος χάρη έχουμε κάποιες εκδηλώσεις όπως η διάσκεψη για τη Συρία που έχει γίνει ετήσια ακριβώς για να ε, συλλέξουμε περισσότερη στήριξη και να ζητήσουμε περισσότερες οικονομικές εισφορές από τα κράτη-μέλη. Τώρα, φυσικά πολλές φορές ε, έχει τεθεί το ερώτημά σας ε, για το θέμα της Βόρειας Συρίας, αλλά δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των επικεφαλής, ε, ότι δεν ε, θα ε, προσφέρουμε στήριξη στην νοικοδόμηση αν δεν είναι η κατάσταση στη Συρία ασφαλής. Δηλαδή μιλάμε και για εκούσιες επιστροφές από οπουδήποτε και αν είναι. Σας ευχαριστώ. Αν ο κ. Σουρέλη θέλει να προσθέσει κάτι από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Budget, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν εξαντλητικό ο συνάδελφο Φοβόφσκι. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Νομίζω πολύ καλά εξήγησε τη φύση την ίδια τη πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ένα νέο μέσο που προτείνουμε που θα συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα έτσι με τα λόγου γνώσεως και που να έχει βάση αν δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις για το μέσο αυτό. Ε, δεύτερο, αναφέρθηκε ο συνάδελφός μου, η παράταση του Ταμείου Μαντάτ κατά ένα έτος έχει ένα αντίκτυπο που έχει ήδη συμπεριληφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή δεν θα επηρεάσει ε, την πρόταση της Επιτροπής και τον προϋπολογισμό μια τέτοια απόφαση. Και ένα τρίτο έτσι, γενικό σχόλιο και υπενθύμηση ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα η Επιτροπή σας ε, παίρνετε ε, ε, αναφορά, η Επιτροπή Προπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου βλέπετε αναλυτικά κατά καταπίστευμα τις λεπτομέρειες και των συνεισφορών ανακράτος μέλος και τα λοιπά. Αναλυτική αναφορά με πληροφορίες και λεπτομέρειες, ό,τι χρειάζεστε για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρέλ. Σχόλια. Έχετε άλλα τα μέλη της Επιτροπής των Επιτροπών. Αν όχι, μπορούμε να κηρύξουμε το πέρας της συνεδρίασης και εξ ονόματο του κυρίου Βοητσεχόφσκη. Οι συντονιστές των δύο επιτροπών θα εκπονήσουν σύσταση, η οποία θα αποσταλεί στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η σύσταση αυτή θα περιγράφει τα συμπεράσματα της σημερινής ανταλλαγής απόψεων και θα συνυπογράφεται από τους δύο προέδρους των Επιτροπών. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα ενημερώσει την Ολομέλεια και θα αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου θα διαβιβάζεται η επίσημη θέση του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και για τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θα σας δώσω ραντεβού για αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Το σημαντικότερο. Έχουμε τώρα μία μικρή δεξίωση. Βιαστείτε να προλάβετε.